Siamo pronti? Prendete posto. Buongiorno Καλημέρα σε όλους. Αρχίζουμε την Επιτροπή μας και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρξουν και παρατηρήσεις πριν από το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά της 12ης Μαρτίου και της 16ης Απριλίου εγκρίνονται. Σας πληροφορώ, πληροφορώ δηλαδή όλη την Επιτροπή, ότι αύριο μαζί με τους συντονιστές θα συναντηθούμε με τον Επίτροπο Τσόλος για να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την επιτροπολογία, την πρώην επιτροπολογία, η οποία θα γίνει βασική πράξη πλέον ή συμπληρωματική πράξη. Ελπίζω να, βρω, να βρούμε συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα, ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να παίξει το ρόλο του ως νομοθέτηση, έτσι όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Επιπλέον να σας πω ότι θα έχουμε και ένα workshop λέει ο πρόεδρος, μια συνάντηση στις 10 Μαΐου και μία έκτακτη συνεδρίαση στις 18 Μαΐου, στις 7 το βράδυ στο Στρασβούργο αυτά, για να εξετάσουμε τις πολυάριθμες τροπολογίες ε, στην έκθεση του George Lyon για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013. Να αρχίσουμε τώρα με ε, την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τζον Ντάι, ο οποίος είναι επίτροπος ε, για, τους, ε, για την προστασία των καταναλωτών. Σε καλωσορίζω αγαπητέ Τζον. Όλοι μας οι βουλευτές ενδιαφέρονται να μάθουν ποιο είναι το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν στο μέλλον για τα υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά ζητήματα και την ευημερία των ζώων και την τροφιμική ασφάλεια. Λοιπόν, έχεις το λόγο. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είναι μεγάλη η χαρά μου σήμερα που βρίσκομαι κοντά σας σε μια πρώτη ευκαιρία να σας ενημερώσω για σημαντικά θέματα ενδιαφέροντος της Επιτροπής σας. Θα μπορέσω βέβαια και να απαντήσω και στις ερωτήσεις που ίσως θέλετε να μου υποβάλλετε. Η γεωργία και η βιομηχανία τροφίμου είναι πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι ο μεγαλύτερος μεταποιητής και ο μεγαλύτερος εργοδότης. Γι' αυτό το τομέας αυτός έχει θεμελιώδη σημασία. Τα λέω αυτά για να τονίσω τη σημαντική συμβολή της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμου και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων ε, του 2020. Εγώ θα ρίξω φως στους ε, στόχους της Γενικής μου Διεύθυνσης. Όπως προκύπτει από την τρέχουσα κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται, η φύση χρειάζεται προστασία απέναντι στους οργανισμούς που, την, ε, που είναι επιβλαβείς. Το ίδιο και για ε, νόσους ασθένειες των φυτών οι οποίες προκύπτουν από τις κλιματικές αλλαγές. Στόχος μου είναι μέχρι το 2012 να υποβάλω νέα στρατηγική για την προστασία της υγείας των φυτών. Επίσης, σχετικά με την εφαρμογή του νέου ε, νομικού πλαισίου για την προστασία των φυτικών προϊόντων. Εδώ υπάρχει σαφές κίνητρο για να προβεί σε καινοτομίε η βιομηχανία ζυζανιοκτώνων και να προσφέρει στην αγορά ασφαλέστερα προϊόντα που θα ωφελήσουν του πάντε. Τα νέα προϊόντα στο μέλλον θα φθάνουν στι αγορέ συντομότερα λόγω των πιο σφιχτών προθεσμιών για τις εγκρίσεις, ανοίγοντα έτσι το δρόμο σε ταχύτερη και ομαλότερη πρόσβαση των γεωργών. Σχετικά τώρα με τους, μη, με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, όπως θα γνωρίζετε, υπάρχει και μια δράση μέσα στο πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε μέχρι τον Ιούνιο να υποβάλει συγκεκριμένη πρωτοβουλία για το πώ θα μπορέσουν οι χώρε μέλη να έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν εάν θα εγκρίνουν ή όχι την καλλιέργεια ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφο του. Ανταποκρινόμενοι έτσι στι θέσει του Πρόεδρου Βαρόσο και στι ε, πολιτικέ θέσει που ε, διατύπωσε πριν από την ε, σύνθεση τη Κομισιόν. Ήδη τον Ιανουάριο ανέλαβα υποχρέωση να υποβάλω σχετική έκθεση μέχρι τέλους του έτους. Και ο τομέας αυτός περιλαμβάνεται και μέσα στο πρόγραμμα εργασιών. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν, επί του παρόντος, προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους, ούτως ώστε να έχουν μια συνολική επισκόπηση. Με την ευκαιρία θα εξηγήσω τις θέσεις μου σχετικά με το μέγα θέμα της καινοτομίας και της επιστημονικής πρόοδου. Εγώ είμαι υπέρ της καινοτομίας και δεσμεύομαι να βελτιστοποιήσω τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει, αλλά και βέβαια με οποιοδήποτε κόστος. Θα ακολουθήσω πολιτική υπεύθυνη καινοτομία, όπου θα ενισχύεται κάθε προσπάθεια πρόοδου, αλλά ταυτόχρονα με πλήρη εξέταση κινδύνων και ασφάλειας. Ήδη αναφέρθηκα στις ε, πιο αυστηρή, στην πιο αυστηρή νομοθεσία σχετικά με τις εγκρίσεις νέων προϊόντων. Χρειαζόμαστε πιο ανοιχτή και συνολική συζήτηση με συμμετοχή και της βιομηχανίας σχετικά με τις ωφέλειες που θα προκύψουν για υπέρ των πολιτών από τα διάφορα καινούργια καινοτόμα προϊόντα. Όσο θα γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση το 2007 για μια νέα στρατηγική προστασία των ζώων θεωρώντα ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την καταστολή. Η στρατηγική αυτή ακολουθήθηκε το Σεπτέμβριο 2008 από την έγκριση συγκεκριμένου σχεδίου δράσεων, από τι οποίε οι περισσότερε δράσει έχουν αρχίσει να ε, λειτουργούν και ορισμένε έχουν αποδώσει καρπούς. Ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο τη στρατηγικής αυτή, εγώ πρόκειται να κάνω ε, σχετική πρόταση νόμου στι αρχέ του επόμενου έτου. Θα πρέπει να μην λησμονούμε την σχέση μεταξύ των κανόνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των διεθνών κανόνων η νομοθεσία μας συμμορφούται γενικά με τους κανόνες της ε, Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Προστασία των Ζώων. Ορισμένοι από τους κανόνες μας μάλιστα βαίνουν και μακρύτερα. Εμείς θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε δικαίωμα ε, να διατηρεί υψηλά επίπεδα ή υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας του κοινού και προστασίας των ζώων όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η πρώτη δράση 2006-2010 λύγει φέτος και αξιολόγηση των επιτευγμάτων της βρίσκεται ήδη στο, στη φάση της συντάξεως και θα δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο. Ιδιαίτερη προσοχή έχουμε δώσει στην αξιολόγηση των δεδομένων του κόστους, σχετικά δηλαδή με την τήρηση υψηλών γραφών προστασία των ζώων. Σχετικά με αυτό και με τις συστάσεις της πολύ χρήσιμης Έκθεση Πούλσεν τη ε, επιτροπή σα. Εμεί βασιζόμενοι λοιπόν σε αυτό φτιάχνουμε μια νέα στρατηγική η οποία θα είναι ολιστική και θα αναφέρεται στις, ως όλες τις πολιτικές ευημερία των ζώων για τα επόμενα χρόνια. Άλλο θέμα τώρα ευημερία το οποίο ήταν δύσκολο στο παρελθόν. Η προστασία δηλαδή των ζώων κατά τη διάρκεια τη μεταφορά των. Εδώ έχει αναλάβει την υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση το δεύτερο εξάμεινο του επομένου έτους και βασισμένη σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα του θέματος. Και βέβαια και σχετικά με την τήρηση και επιβολή των νησιώτων κανόνων. Για άλλα θέματα τώρα, τα οποία έχουν σχέση με την ευημερία ε, των ζώων, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσεως, θα σας αναφέρω τη σχετική ε, προσπάθεια επισήμανσης, με ε, το labeling δηλαδή των δεν θα πούμε εμείς στον κόσμο τι θα τρώει, αλλά έχουμε καθήκον να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς τρώει. Τον προηγούμενο Οκτώβρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκθεση που περιλάμβανε ε, πλήωνα θέματα σχετικά με την επισήμανση των ζώων και επίσης κέντρα αναφοράς για τις, για τις σχετικές αυτές ε, ε, προσπάθειες. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ιδέες και μέσα στην έκθεση για θέματα τώρα ασφάλειας των τροφίμων και προστασίας των ζώων, η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος και πραγματικά βρίσκεται σε υψηλό, επίπεδο παγκοσμίω. Έχουμε και τεράστιο δυναμικό. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό αυτό με την ευρύτερη έννοια για να ανοίξουμε ε, αγορές, να ανοίξουμε ευκαιρίες στις αγορές. Είναι εξαιρετικό το εμπορικό μα σήμα, α το πούμε έτσι, α το εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο. Θα πούμε λοιπόν καθαρά ότι τα εισαγόμενα προϊόντα πρέ, οφείλουν να τηρούν τις προδιαφέ ασφαλείας μας και ε, να είναι ανάλογα με αυτά που παράγονται στην Ευρώπη. Ωστόσο, για να εξετάσουμε και το θέμα της ανταγωνιστικότητας, εγώ θα υποβάλω έκθεση μέχρι τέλος του 2010 για ε, τα θέματα των εισαγόμενων προϊόντων. Θα έρθω σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, γιατί αυτό βεβαίω είναι θέμα το οποίο ενισχύει πολλού. Ωστόσο, πάντοτε η κόκκινη γραμμή θα είναι ότι πρέπει να συνεχίσετε να παράγετε τρόφιμο ασφαλές και για όλους. Για τα TSC, νομίζω ότι φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο όπου μπορούμε να προχωρήσουμε στη λήψη και νέων μέτρων χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Γι' αυτό ζήτησα από τι υπηρεσίε μου να φτιάξω ένα ε, οδικό χάρτη για το TSC για την περίοδο 2010 2015. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να εγκριθεί ήδη τον Ιούνιο και θα διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο για να αρχίσει η συζήτηση. για τη σπογγόδια κεφαλοπάθεια. Οι γεωργοί, παραγωγή τροφίμων και νομοθέτες μπορούν να υπερήφανοι για τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για την προσφορά στους καταναλωτές ασφαλών και φθηνών τροφίμων. Η επιτυχία αυτή μπορεί να συνεχιστεί μονάχα εφόσον τα μέτρα που ήδη έχουν εγκριθεί συνεχίσουν να εφαρμόζονται και να τηρούνται ε, στόχο την αύξηση Τη αξιοπιστία του ρυθμιστικού πλαισίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, αυτή είναι μια σύντομη επισκόπηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που πήρα από το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπή και πρόσθεσα ορισμένα άλλα. Ευχαρίστω τώρα θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Έχουν ζητήσει πολλοί βουλευτέ το λόγο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως τη συζήτηση και φυσικά σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο γιατί έχουμε και μια βεβαρημένη μερισιά διάταξη. Η κυρία Ελίζαπετ Αγγέλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε για την έλευσή σας εδώ. Ευχαριστώ και για τις δηλώσεις σας. Στις οποίες αναφερθήκατε σε θέματα που και μας μας απασχολούν, όχι μόνο στην εργασία μας αλλά και στις σκέψεις μας. Μια πρώτη ερώτηση. Όταν λέτε 2012 νέα στρατηγή προστασίας των φυτών, μόλις εγκρίναμε την δέσμη μέτρων για την προστασία των φυτών. Γιατί τώρα βιάζεστε τόσο, τόσο σύντομα, δηλαδή έρχεστε πάλι να διατυπώσετε νέα στρατηγική. Το άλλο μεγάλο θέμα ήταν η προστασία των ζώων. Εγώ είχα αναλάβει την σύνταξη της εκθέσεως του Κοινοβουλίου για τη στρατηγική, η οποία λύγει τώρα, 2006 δηλαδή μέχρι 2010. Και, και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επιτύχαμε νέα πράγματα με την συζήτηση αυτή και με την στρατηγική αυτή δώσαμε μια όθηση προς την βελτίωση της ε, προστασίας των ζώων σε όλη την Ευρώπη. Λέτε τώρα ότι θέλετε πιο μακροπρόθεσμα να ψηφιστεί ευρωπαϊκός νόμος για την προστασία των ζώων. Υποθέτω ότι ε, μεγάλο μέρος της Επιτροπής Γεωργίας θα ε, συμφωνήσει σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση και την ενιαία αγορά που χτίζουμε μαζί. Αλλά και για ζώα, δηλαδή ζώα της αγροτικής εκμετάλλευσης, αλλά και πειραματόζωα κτλ. Βάλτε μέσα σε αυτή τη ρύθμιση και άλλα ζώα, όπως για παράδειγμα αδέσποτα σκυλιά και γάτες. Όταν λοιπόν μιλούμε για προστασία των ζώων, ας μιλήσουμε για το σύνολο των ζώων που χρειάζονται προστασία. Για την συζήτηση τώρα σχετικά με την στρατηγική που θα έρθει μετά και η κυρία Πόλσεν θα συζητήσει και το θέμα αυτό στην έκθεσή της και εγώ τη συγχαίρω πάντως για τη μέχρι τώρα πορεία της εκθεσεώς της. Ωστόσο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να τεθεί και το εξής ερώτημα. Από τη στρατηγική στην οποία αναφερθήκατε τι έχει εφαρμοστεί, πού έχουμε φτάσει μέχρι τώρα ενώ τη μεταφορά των ζώων. Σε ποιες χώρες γίνεται κάτι σε ποιες χώρες χρειάζεται ακόμα να προχωρήσουν τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για τους κανονισμούς ε, εκτροφής και διατήρησης των ζώων. Τώρα, ευρεσιτεχνίες για ε, βιολογικά προϊόντα και για την κλωνοποίηση. Είπατε ότι θα υποβάλλετε έκθεση μέχρι τον Ιανουάριο. Ε, σημαντικό θέμα αυτό, το ίδιο σημαντικό και βεβαίως μπορεί κανείς να το εξετάσει και, στην ίδια, και στο ίδιο πλαίσιο οι δύο ε, ευρεσιτεχνίε, αν μπορώ να πω έτσι. Είναι λοιπόν σημαντικό θέμα και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ευχαριστώ, Ελίζαμπεθ. Μισελ Νταντέν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για τον οδικό χάρτη που μόλις μας παρουσιάσατε. Νομίζω ότι είναι πλήρης, σαφής ε, και περιλαμβάνει ένα καλό χρονοδιάγραμμα, μας έχετε δώσει πολλά ραντεβού, θα είμαστε πιστοί. Θα ήθελα όμως να επανέλθω σε ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκατε. Πρόκειται για το αυξανόμενο κόστος, το υψηλό κόστος των ε, μέσων προστασίας που επιβαλούμε για την ε, χειρουργική προστασία στην Ευρώπη. Από ό,τι κατάλαβα είπατε ότι θα γίνει αξιολόγηση του κόστου αυτού. Δεν σημείωσε το χρονοδιάγραμμα αυτή τη αξιολόγηση. Νομίζω ότι είναι όμω ε, στο πλαίσιο τη συζήτηση που ξεκινάμε για την ε, κοινή αγροτική πολιτική και των μέλλον τη να δούμε την πτυχή αυτή, γιατί ε, αυτό το αυξανόμενο κόστο θέλουμε να δούμε να αιτιολογούν τι πιστώσει που αφαιρώνουμε στην αγροτική παραγωγή. Και επίση ε, θέλουμε να αναφερθούμε σε μια προβληματική που παρουσιάζεται στην Ευρώπη, νέα προβληματική. Νομίζω όμως ότι θα χρειαστεί σύντομα ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Πρόκειται για τη βιομηχανική ρήπανση. Παντού στην Ευρώπη βλέπουμε σήμερα εκμεταλλεύσεις ε, που φύγονται από ε, την ανακάλυψη παλιάς ρήπανσης, διοξίνες, χάρη, PCB οι γεωργοί είναι θύματα αυτής της κατάστασης και ουσιαστικά δεν υπάρχει ένα πλαίσιο που να επιτρέπει τη συνέχιση της παραγωγής τους. Ενίοτε αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τοπικό επίπεδο. Σκεφτούμε το χάρη τι γίνεται στις περιφέρειες κάποιων εργοστασίων αποτέφρωση ή εκεί όπου έχουμε χημικά εργοστάσια. Εκεί υπάρχουν δεκάδες εκμεταλλεύσεις που θα μπορούσαν να πληγούν και να μην έχουν πρόσβαση στην αγορά για τα προϊόντα τους ε, για πολύ καιρό. Αυτή είναι μια κατάσταση που την συναντάμε και πρέπει να τη θέσουμε σε ένα ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ευχαριστώ μας. Λέω ο κύριος Μποβέ και μετά Σμιτ. Κύριε Πίτροπε, εδώ και κάποιου μήνε τώρα έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σα και είναι αλήθεια ότι ξεκινήσατε ε, με ιδιαίτερη ορμή, δεχόμενο ε, και προωθώντα ε, την έγκριση των γενετικά, τροπο, της γενετικά τροποποιημένης πατάτας. Και έτσι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Ευρωπαίοι καλλιεργητέ πραγματικά εξεπλάγησαν. Ήταν ένα σοκ αυτό και ε, κανείς ε, ε, ε, δεν καταλαβαίνει γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η αξιολόγηση της ΕΦΣΑ ε, που έχει ζητηθεί εδώ και ένα-δύο χρόνια και πώς μπορούμε να δεκτούμε συστηματικά ακόμη και σήμερα να δίνουμε έγκριση ενώ ξέρουμε ότι ο οργανισμός αξιολόγησης ε, ουσιαστικά δεν είναι στο ύψος των όσων διακυβεύονται σήμερα σε επιστημονικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο σήμερα. Ε, μας είπατε ότι για τον Ιούλιο θα προτείνετε νέα νομοθεσία που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη μέσω της επικουρικότητας ε, να δεκτούν ή να αρνηθούν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η κατάσταση θα καταστεί πολύπλοκη στο μέτρο που άλλα κράτη θα δεχτούν ή θα απαγορεύσουν ε, τους γενετικα τροπομενους οργανισμους το προβλημα ειναι οτι αυτη η ομικρών. Αυτό δεν διευκολύνει ε, το να έχουμε μια κοινή αγορά. Μπορούμε να έχουμε και προβλήματα επιμόλυνσης με τη γύρη και τα λοιπά. Μπορούν να περάσουν από τη μία χώρα στην άλλη. Και μάλιστα το να διαχειριστείτε αυτό το θέμα με αυτόν τον τρόπο δεν είναι συνεπές. Και υπάρχει και ένα τρίτο πρόβλημα που τίθεται έχει να κάνει με την ε, ε με τον ΠΟΕ. Δηλαδή θα βρεθούμε σε μια κατάσταση κάποια κράτη-μέλη που έχουν αρνηθεί τους γενετικά τροπομένους οργανισμούς να μπορούν να δεχτούν επίθεση σε ένα πάνελ ε, του ΠΟΕ. Γιατί θα έρχεται αυτό σε αντίθεση με τους κανόνες που θα έχει δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτι άλλο ε, σε ό,τι αφορά τους τύπους, τη μορφή. Δηλαδή δεν είναι αποδεκτό σήμερα η συζήτηση συζήτηση αυτή γίνεται παρά των Κομισιών, τα κράτη-μέλη και συμμετέχουν. Δηλαδή εδώ θέλουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολίτες να συμμετέχουν. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να συζητήσει το θέμα αυτό. Δεν είναι λογικό η συζήτηση αυτή να γίνεται μόνο στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν και να περιοριστεί εκεί. Θέλω μια σαφή απάντηση για αυτό το θέμα λοιπόν. Δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα αφορά την διατροφή εδώ και χρόνια εμείς ε, αγωνιζόμαστε και η Κομισιόν σε όλες τις εκθέσεις μας μιλά για την ποιότητα μόνο σε ένα θέμα κεντρικής σημασίας. Προωθεί την ποιότητα. Σήμερα όμως βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας πρότασης που μπορούμε να την ονομάσουμε junk food. Πρόκειται ε, την πρόταση που επιτρέπει ε, να έχουμε έναν επεξεργασμένο κρέας. Δηλαδή θα επιτρέψουμε προϊόντα όπως το Fibrimex να μπει ε, στη διατροφική αλυσίδα, δηλαδή να έχουμε πολλαπλά κομμάτια κρέας και να μας δίνεται η εντύπωση ότι έχουμε ένα τεμάχιο κρέας ενώ θα είναι πολλαπλά ε, τεμάχια όπως έχουμε παίρνει το τον κορδόν μπλε του κοτόπουλου. Ε, δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο σε μια πολιτική ποιότητα και γι' αυτό παροτρύνω τώρα τους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια να ψηφίσουν προς την ίδια κατεύθυνση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος η οποία ψήφισε σε μαζικά υπέρ τη απαγόρευση του προϊόντος αυτού. Θα ήθελα μια απάντηση λοιπόν και για αυτό το ζήτημα από εσά. Κύριο Σμιτ, παρακαλώ. Uh, uh, uh, Καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε. Δύο θέματα. Μεταφορά των ζώων και τα trans τα ε, αυτά. Όπω είπε και η κυρία Γέγλε, γνωρίζουμε στην Επιτροπή μας ότι υπάρχουν θέματα συμμόρφωσης ε, των χωρών μελών ε, στους κανόνες προστασίας ε, των ζώων ή μεταφορά των και το λαμβάνουμε υπόψη. Μου διαφαίνεται κάποια αλλαγή στην στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλήσατε για καλύτερη επιβολή των κανόνων. Θα γνωρίζετε ότι στη Σκωτία την εκλογική μου περιφέρεια υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι ίσως με την ευκαιρία αυτή θα επιβληθούν νέοι κανόνες ενώ τώρα μόλις έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε τους ισίοντες. Αν μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε λοιπόν ότι θα ρίξετε ιδιαίτερο βάρος στην ε, επιβολή των ισχυρων κανόνων. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα καλό δεκτό από εμά. Για τα trans τώρα, όπως είπε και ο Ζωζέ Μποβέ, υπάρχει γραπτή διακήρυξη από διάφορους ευρωβουλευτές η οποία θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει τα ε, λύπη αυτά από ε, τη χρήση τους δηλαδή στην ε, ε, ανθρώπινη διατροφή. Ίσως μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ελπίζουμε να υποστηριχθούμε από πολλούς ευρωβουλευτές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην διακήρυξη μας αυτή. Ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Η κυρία Πόλσεν. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Έχω την εντύπωση ότι εδώ λειτουργώ σαν παπαγάλος που εδώ και 34 χρόνια επαναλαμβάνει τέτοια πράγματα. Αλλά να σας πω, είμαι μεγάλη γυναίκα και πρέπει τελικά μάλλον να δεκτώ ότι είμαι και παπαγάλος. Ό,τι αφορά τώρα την υγεία των ζώων και σε συνδυασμό με τη δημόσια υγεία. Σήμερα υπάρχει ένα ζωτικό θέμα αφορά την ε, αντίσταση, την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Ξέρω ότι ψηφίσαμε την ε, απαγόρευση της χρήσης αντιβιωτικών ως ε, συστατικό για την ε, ανάπτυξη των ζώων. Και τώρα έχουμε μια συνολική εικόνα σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα αντιβιωτικά στη δημόσια υγεία, αλλά χρειαζόμαστε και μια παρόμοια μελέτη για να γνωρίζουμε σε ποιους τομείς, για ποιες ασθένειες, για ποια ζώα χρησιμοποιούνται τα αντιβιωτικά σήμερα. Γιατί τα αντιβιωτικά είναι σημαντικά και για τα ζώα αλλά και για τον άνθρωπο. Να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά. Ένα ζώο το οποίο φέρει μεταδοτική νόσο, σοβαρή, Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα αντιβιωτικά με τον ίδιο τρόπο όπως και για τον άνθρωπο. Όμως δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση των φαρμάκων αυτών. Κάτι ακόμη. Θα τολμήσουμε να αναφερθούμε στη συζήτηση για τις νέες βιολογικές τεχνολογίες η τεχνολογία των γενετικών τροπομενων οργανισμών, θα την αναφέρουμε, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και κάθε σκεπτικισμό. Σήμερα η επιστήμη μας επιτρέπει το γενετικό χειρισμό, τη γενετική χειραγώγηση με μεθόδους που δεν λέγονται γενετικά τροποποιημένες. Δεν έχω χρόνο τώρα να αναφερθώ λεπτομερώς σε όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να γίνουν κάποια σεμινάρια στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να έλθουν εδώ κάποιοι επιστήμονες ε, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να μελετήσουμε εις βάθος την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών και να δούμε πώς ε, μπορούμε να νομοθετήσουμε και πώς να αποκαλέσουμε τις τεχνολογίες αυτές. Γιατί δεν γνωρίζουμε καθόλου ε, το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν εγώ ζητώ να έχουμε όλο ένα και περισσότερες γνώσεις. Ευχαριστώ κυρία Πόλσον Μαγκίνες. Thank Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Άκουσα και τις προκαταρκτικές σας παρατηρήσεις σχετικά με τη σημασία της Γεωργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το 2020, αν και αυτό το είπατε κάπως αργότερα. θα τα συζητήσετε αυτά σήμερα το απόγευμα στην Κομισιόν σχετικά με συζητήσεις που θα αρχίσετε με τις χώρες Mercosur σχετικά με διμερείς συμφωνίες που θα έχουν σημαντική επιρροή στην ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία και κυρίως τον τομέα της πτηνοτροφίας και του βόλου κρέατος. Η κατάσταση του βόλου κρέατος της Βραζιλίας είναι γνωστή και μας ανησυχεί. Θα αρχίσουν πάλι αυτές οι συζητήσεις λοιπόν. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας, της προστασίας και της ευημερίας των ζώων, αυτά είναι καλά. Αλλά μήπως αυτές οι συζητήσεις πρέπει να γίνουν πριν από τις συζητήσεις που θα γίνουν στον ΠΟΕ. Θα ήθελα να κάνετε κάποια σχόλια και θα ήθελα να μεταφέρετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχόλια των Ευρωπαίων Γεωργών. Ιδίω σε μια περίοδο όπου μειώνεται σημαντικά το εισόδημά τους. Δεύτερο, μιλήσατε για, τα, ε, για τις υψηλές προδιαγραφές που απολαμβάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας απασχολεί πολύ. Δεν κάνετε αρκετά όμως για να προστατεύσετε τους Ευρωπαίους αγρότες απέναντι στις εισαγωγές από τρίτες χώρες όπου έχουν διαφορετικές προδιαγραφές. Ωραία είναι τα λόγια, αλλά υπάρχει και η ιδέα της ισότητας και της ισοδυναμίας. Εάν επιβάλλεται πολύ ψηλέ προδιαγραφέ που αυξάνουν το κόστο παραγωγή των Ευρωπαίων αγροτών, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούν τότε να ανταγωνιστούν τι εισαγωγέ από τρίτε χώρε, όπου έχουν άλλε προδιαγραφέ και κατά τη γνώμη μου ε, μειωμένε. Τώρα για τα GMO, για του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει εδώ στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα GMO. Α αναγνωρίσουμε τι πραγματικότητε, τουλάχιστον για τι ζωοτροφέ. Και έρχομαι στο θέμα της ανοχής για τις ζωοτροφές. Και ίσως μπορείτε να μου απαντήσετε και γραπτός για να μου ε, μιλήσετε για τον τομέα ε, του τροφίμου και για την ανοχή εκεί, τις ανοχές εκεί ε, απέναντι στους GMO. Είναι θέματα, όπως είπα, πραγματικότητα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, για τις μεταφορές των ζώων. Εγώ υποστηρίζω την ιδέα της καλύτερης επιβολής μην μα ζητείτε όμω να συμφωνήσουμε να θεσπιστούν νέοι κανόνε όταν ακόμη δεν εφαρμόζονται οι παλαιοί. Και κυρίω σχετικά με τη μεταφορά αλόγων, που είναι θέμα ευημερία των ζώων αυτών και βεβαίω η μεταφορά του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και τώρα σε ό,τι αφορά την επισήμανση, το labeling, αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα των ε, αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ό,τι και να κάνουμε εδώ, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ουσία παίζουμε δεύτερο βιολί απέναντι στο τι κάνει το λιανεμπόριο εφόσον έχουμε τις υψηλές αυτές προδιαγραφές, πρέπει να έχουμε και πληρωμές υπέρ των παραγωγών. Δεν νομίζουμε ότι αυτό θα γίνει μέσω ε, δημοσίων χρημάτων και πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη και για τη μεταρρύθμιση του 2013. Όντω έχουμε ένα εξαιρετικό εξαιρετική ποιότητα εμπορικό ΣΥΠΑ ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμω ακριβό και χρειάζεται και πληρώνεται και το πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εξυψωθούν και τα παγκόσμια στάνταρτ και να φτάσουν στα δικά μας και όχι να υπάρχει ανταγωνισμός ε, προδιαγραφών. Και για τη σπογκώδη κεφαλοπάθεια, μετά από, την, ε, από τον Ιούνιο είπατε ότι θα έκθεση, τα θέματα είναι πολλά και πράγματι βαθιά ακούσαμε από τα ε, φθηνά τρόφιμα, από τα junk food δηλαδή μέχρι την κλωνοποίηση. Είναι όμως σημαντικό το θέμα της προστασίας των αγροτών. Χρειαζόμαστε να υπάρχουν οι αγρότες και, και αυτοί πρέπει να ζήσουν. Grazie onorevole McGuinness. Adesso George Lyon, poi Luis Santos e poi diamo la possibilità a Commissione. Ο George Lyons και μετά ο Κάπουλα Σάντο, και μετά θα απαντήσει ο Επίτροπο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Επίτροπο που ε, παρευρίσκεται εδώ και απευθύνθηκε σε εμά. Ε, αναφέρθηκαν αρκετά θέματα, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον οδικό χάρτη για τι μεταδεδομένε και κεφαλοπάθειε που θα εκδώσετε τον Ιούνιο. Θα δούμε κάποια πρόοδο, δηλαδή να τεθεί ένα τέλο στι δοκιμέ, καθώ ε, έχουμε πολύ χαμηλά κρούσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότερε από αυτέ ε, τι περιπτώσει, περισσότερα από αυτά τα κρούσματα ανακαλύφθηκαν μετά το θάνατο. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά δεν εντάσσονται στο διατροφική λυσίδα. Επίση, το θέμα τη μεταφορά των ζώων τέθηκε από αρκετού συναδέλφου. Είπατε ότι το επόμενο εξάμεινο ή το, δεύτερο εξάμεινο του 2011 θα εκδώσετε μία έκθεση. Θα δοθεί έμφαση στην επιβολή της νομοθεσίας ε, παρά θα έχουμε νέα νομοθεσία για τη μεταφορά, γιατί αυτό το θέμα προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία και στην Ευρώπη αλλά και στη Σκωτία. Τρίτον, ε, υποσχεθήκατε μία έκθεση για τις ε, εισαγωγές. Αυτό είναι ένα θέμα που το συζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν την Επιτροπή και σίγουρα πριν και τη δική μου θητεία. Εξακολουθεί να μας ενσυχεί ότι ορισμένες ε, από τις εκθέσεις ΦΑΟ δείχνουν καλή πρόοδο σε σχέση με το βόλιο κρέας από τη Βραζιλία, αλλά υπάρχουν ανησυχητικά θέματα στην έκθεση, προβλήματα με τα καθεστώτα εποπτείας, με την χνησιμότητα μπορείτε να μα πείτε αν είστε ικανοποιημένο με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ή αν θα πρέπει να, ληφθεί περαιτέρω, να ληφθούν περαιτέρω δράσεις σε σχέση με το να βελτιώσουμε την ειχνημεσιμότητα για το ε, βόλιο κρέα από τη Βραζιλία και σε σχέση με τη βελτίωση των καθεστώτων αποκτία. Ευχαριστώ, Λουίς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας. Ε, κύριε Επίτροπε, δύο ερωτήσεις. Ε, το ένα θέμα έχει να κάνει με το πραγματικό έλεγχο των υγειονομικών και φυτογειονομικών μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από το θέμα της διαφύλαξης της υγείας των ζώων και των ανθρώπων, όπως ξέρετε, είναι το έσχατο σύνορο οι κανόνες αυτές. Ε, σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε, για την έκθεση που θα παρουσιάσετε, αλλά όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, μας ανησυχεί περισσότερο η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της υφιστόμενη νομοθεσίας παρά η ενδεχόμενη εκπόνηση νέας νομοθεσίας Σα ε, εγώ μπορώ να σας εγγυηθώ ότι πηγαίνω έρχομαι μεταξύ Βρυξελών και Πορτογαλίας και βλέπω ότι υπάρχει δυσκολία ε, των αρχών της Πορτογαλίας να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στο θέμα αυτό. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε στην έκθεση αυτή θα συμπεριληφθεί και κάποια αξιολόγηση για τη συγκεκριμένη εφαρμογή αυτών των κανόνων στα διάφορα κράτη-μέλη ή αν ε, μπορείτε να μας δώσετε ήδη κάποια αξιολόγηση. Δεύτερη ε, ερώτηση έχει ε, να κάνει με την ασθένεια των ε, πεύκων. Όπως ε, ξέρετε, το, 80, το 2000, από το στο 2000, στην Πορτογαλία είχαμε την νόσο των πεύκων να έρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείες, από ε, ξυλία που εισήχθη από τις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, και ξέρετε ε, δεν ήταν δυνατό να εξαλείψουμε την όσο αυτή και δυστυχώς υπήρξε και εξάπλωση και σε άλλα κρατημέλη. Θα θέλω να μου πείτε υπάρχει κάποιο σχέδιο πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να προλαμβάνουμε την διάδοση της νόσου αυτής η οποία μπορεί να έχει πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις για τα δάση στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι τώρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Επίτροπο για να απαντήσει σε αυτή την πρώτη ομάδα ερωτήσεων και κατόπιν έχουμε και οκτώ μέλη ακόμη που έχουν ζητήσει το λόγο. Νομίζω όμως ε, ότι καλό θα ήταν να δώσω σε εσά το λόγο. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας μου δίνεται και την ευκαιρία να επεκταθώ και σε κάποια ζητήματα μέσω των ερωτήσεων που ακούστηκαν. Ε, πρόσφατα, εμείς ε, με μια νομοθεσία για τα φυτοφάρμακα, για τα φυτοφάρμακα προϊόντα και όχι για την ε, ευημερία των ζώων. Έτσι, η νέα μας στρατηγική θα επικεντρώνεται περισσότερο στην ευημερία των ζώων και θα βασιστούμε σε μεγάλο βαθμό στα συμπεράσματα που ε, έχουμε στην έκθεση Πόλσεν, την οποία έχουμε δεκτεί και τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής να σας πω ότι συνάδουν και με τη δική μας συλλογιστική. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε λοιπόν την κυρία Πόλσεν για τη συνεισφορά της στον τομέα αυτό και φυσικά όλοι έχουμε να κερδίσουμε από τη μεγάλη της εμπειρία στον τομέα. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ζώων, ε, αυτό το θέμα τέθηκε από πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εγώ θεωρώ ότι πριν ε, να ξεκινήσουμε με την εκπόνηση νέας νομοθεσίας πρέπει να αναλύσουμε το καθεστώς της σημερινής νομοθεσίας των φυστάμενων κανονισμών γιατί η ανάδραση που λαμβάνω, το feedback που λαμβάνω είναι ότι η φυστάμενη νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στο κατάλληλο επίπεδο στα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στο εξή. Να ε, προωθήσουμε την επιβολή της νομοθεσίας, την εφαρμογή της νομοθεσίας και φυσικά τα μέσα του 2011 θα εκπονηθεί και η έκθεση που σας ανέφερα δεν θα επικεντρώνεται μόνο στην επιβολή της νομοθεσίας αλλά θα εξετάζεται και η δυνατότητα να δούμε αν ε, δηλαδή υπάρχουν νέε πληροφορίες επί νέων πρακτικών που θα έχουν αναπτυχθεί και δυνάμει αυτού να δούμε πώς θα τις ε, ενσωματώσουμε και τις πρακτικές αυτές. Δηλαδή δεν θα προτείνουμε απλώ μια δράση που να αφορά μόνο την επιβολή της νομοθεσίας. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συνολική εικόνα, αλλά θα προσπαθήσουμε καταρχήν να δούμε τι ισχύει ήδη και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί. Επίσης, ε, το feedback που λαμβάνω για το θέμα της μεταφοράς των ζώων και της επισήμανσης της χώρας προέλευσης. Ε, δηλαδή, τα ζώα μεταφέρονται τεράστιες αποστάσεις ε, για να γίνει ουσιαστικά τελικά μια δήλωση ότι έχει σφαγιαστεί το ζώο σε μια συγκεκριμένη χώρα και όχι σε μια άλλη. Έτσι, λοιπόν, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πρέπει όλα αυτά να τα δούμε συνολικά και να δούμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε προβλήματα πρακτικά. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των κανόνων και της νομοθεσίας, των κανονισμών. Συμφωνώ και με τις ε, δηλώσεις που ακούστηκαν εδώ, με τα σχόλια που ακούστηκαν εδώ, ότι όλα κοστίζουν, όλα έχουν ένα κόστος. Κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε, κάθε επισήμαση που επιβάλλουμε έχει ένα κόστος είτε αφορά την ευημερία των ζώων, είτε άλλους τομείς. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μία συνολική εικόνα του κόστους ε, του κανονισμού όλης της νομοθεσίας ε, που αφορά τους αγρότες. Ε, δηλαδή ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε και ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τους αγρότες αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα, το υψηλό επίπεδο ποιότητας που έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα ε, στο πλαίσιο της ευημερίας ε, και αναδούμε πώς ε, όλοι οι κανονισμοί για την ευημερία των ζώων εφαρμόζονται και ποια είναι η σχέση κόστους κόστους-οφέλους αυτών των στοιχείων. Αυτό φυσικά θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να αξιολογήσουμε με ένα πιο έξυπνο τρόπο θα έλεγα, με πιο ευφυή τρόπο, τα νέα σύνορα, τα νέα όρια τα οποία πρέπει να φτάσουμε. Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική ρήπανση. Ναι, είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε σε πολλές χώρες. Τα κρατημέλη είναι αρμόδα για να διασφαλίσουν ότι ελέγχεται αυτή η ρήπανση και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία για την κλωνοποίηση. Όπως σας είπα, η Επιτροπή στα τέλη του έτους, μέχρι τα τέλη του έτους, θα παρουσιάσει ένα έγγραφο για την κλωνοποίηση. Αυτό ήδη συζητείται σε διάφορους τομείς, στο Κοινοβούλιο, σε διάφορες επιτροπές. Πραγματικά θα ήθελα να εμπλακούν ενεργά όλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση αυτή και φυσικά παρακολουθούμε και τη διαμορφώση της κοινή γνώμης. για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και σε σχέση με τη γενετικά τροποποιημένη πατάτα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καταρτίστηκε και από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το πώς πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις για τους γαματαφόμικρων. Υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Επομένως, ε, όταν αποφασίζουμε βάση ε, αυτού του πλαισίου, καταλαβαίνω σχόλια ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως να σας πω ότι έχουμε ακολουθήσει στενά αυτό το πλαίσιο σε σχέση με το πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Κομισιόν. Είχαμε συζητήσει σε διάφορες επιτροπές και σε διάφορες συναντήσεις του Συμβουλίου. Όμως δυστυχώς ποτέ δεν κατέληξαν σε μία απόφαση, ούτε θετική ούτε αρνητική. Έτσι λοιπόν ε, η Κομισιόν έπρεπε τελικά να αποφασίσει και μάλιστα δυνάμει πολύ αυστηρών κανόνων. Πρέπει να αποφασίσουμε βάσει της επιστήμης. Και ξέρετε, βάσει των επιστημονικών στοιχείων, και ξέρετε ότι η Κομισιόν έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου προκειμένου να έχει επιστημονική αξιολόγηση δύο και τρει φορέ για όλε τι πτυχέ τη απόφαση αυτή. Πάντα τα, ήταν ε, ευνοϊκά τα αποτελέσματα ε, της επιστημονικής έρευνας και δεν είχε καμία επιλογή η Κομισιόν παρά να εγκρίνει γιατί αν λαμβάναμε μία αντίθετη άποψη, κανένα δεν θα εξυπηρετούσε στο πλαίσιο αυτό. Και τελικά εμείς τι κάνουμε. Θέλουμε να προσδιορίσουμε περαιτέρω τη μεθοδολογία και το νομοθετικό πλαίσιο που χρησιμοποιούμε. Συναντήθηκα με την Group και επέμεινα στη συζήτηση που είχα μαζί του ότι καταρχήν πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δέσμευση για το θέμα του ωφέλους ε, που προκύπτει από τέτοια καινοτομία και πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα καταναλωτές. Πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ε, κατάργηση των ε, γονιδίων ε, που είναι ανθεκτικά στα μικρόβια. Έτσι λοιπόν θα προσφέρουμε όφελος και στους πολίτες όταν θα εξετάζουμε και την εφαρμογή, τη χρήση νέων προϊόντων. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε σχέση με το ενδυνάμιο ωφέλη που μπορεί να προκύψουν και επίσης ε, η παρακολούθηση των αποφάσεων που θα έχουν ε, ληφθεί θα πρέπει να είναι πολύ πιο στενή από τη σήμερα γιατί αυτό θα μας δώσει όχι απλώς την ευκαιρία να ελέγξουμε την ακρίβεια των αξιολογήσεων που θα έχουν ε, υλοποιηθεί αλλά επίσης να προβούμε ε, και σε μελλοντικές εξολογήσεις με περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, την περασμένη εβδομάδα ε, συζήτησα το θέμα αυτό στην επίσκεψή μου και ζήτησα από τις Ηνωμένες να ανταλλάξουν μαζί μας πληροφορίες που έχουν σε σχέση με τη δική του εμπειρία για την καλλιέργεια γενετικά τροπημένων οργανισμών. Αυτοί έχουν πολύ ευρύτερη εμπειρία από εμά, γιατί πιστεύω ότι αν βασιστούμε στα γεγονότα, τότε θα εξελίψουμε ε, αυτό το φόβο, ε, αυτό το σύνδρομο το γνωστό που διέπει αυτή τη συζήτηση μέχρι σήμερα. Και στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζω το σχόλιο της κυρίας Πόλσεν ότι θα πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση για το θέμα αυτό. Και εγώ θα πρέπει να συναντηθώ με τους επιστήμονες, ε, όλοι θα πρέπει να συναντηθούμε με τους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να κατανοήσουμε γιατί πράγμα μιλάμε και τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Γιατί υπάρχουν εξελίξεις στον τομέα αυτό και η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν εμείς αποκοπούμε από τι καινοτομία ε, τελικά η Ευρώπη θα μείνει καθαστηριμένη και δεν είναι κάτι τέτοιο το οποίο επιθυμούμε. Δεν θέλει κάτι τέτοιο η Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά τα λίπητα, trans φυσικά εξετάζουμε όλους ε, τους τομείς, όλα τα στοιχεία που βλέπουν την ανθρώπινη υγεία και για την τελευταία παρέμβαση που ακούστηκε να σας πω ότι η δυναμική μας στο τομέα της υγείας είναι ότι η υγεία των ζώων ε, και η ανθρώπινη υγεία είναι ένα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, Αυτά τα transfats ε, τα εξετάζουμε επίσης στο πλαίσιο των διατάξεων για το διατροφικό μας προφίλ. Ε, Δυστυχώ, η Επιτροπή ΕΝΒΗ έχει καταθέσει κάποιες τροπολογίες που θα εξάλληφαν ε, αυτό το διατροφικό προφίλ για την νομοθεσία των καινοτόμων τροφίμων, για το novel food. Ε, εμείς θεωρούμε ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ε, τι τρώνε, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει και να οθούνται προς το να καταναλώσουν κάποια προϊόντα λόγω ε, κάποιου ωφέλου που μπορεί να προκύψει από τα τρόφιμα αυτά, κάτι που μπορεί να είναι σωστό μεν, αλλά ε, ταυτόχρονα να μην γνωρίζουν ότι υπάρχουν ε, και κάποια αρνητικά συστατικά ε, στο, στα τρόφιμα αυτά. Δηλαδή θα πρέπει να δείχνουμε και τα αρνητικά συστατικά των τροφίμων. Για τους γαματαφόμικρων μικρών επίσης. Ε, θα ήθελα να, να αναφερθώ και σε κάποια άλλα θέματα που έθεσε ο κ. Μποβέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη ρήπανση, την ε, μεταφορά κτλ. Σε ό,τι αφορά τις πατάτες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αναφερθήκατε στην επιμόλυνση, κύριε Μποβέ. Ε, δεν ε, ε, γίνεται γονιμοποίηση μέσω της γύρης, όπως ξέρετε για τις πατάτες και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη πατάτα θα καλλιεργηθεί η πατάτα αυτή κοντά σε εργοστάσια αμύλου που θα τις χρησιμοποιήσουν έτσι λοιπόν δεν μεταφέρονται οι πατάτες αυτές δηλαδή για αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει θέμα μεταφοράς φυσικά θα μπορούσε να υπάρξει το ζήτημα αυτό σε άλλες περιπτώσεις. Όμως ε, φυσικά αυτό θα το λάβουμε υπόψη όταν ε, θα ληφθεί η επιστημονική απόφαση. Θα ληφθεί υπόψη ως ένας παράγοντας ασφάλειας. Κύριε Πόλσεν, αναφέρετε την ε, ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Ναι, συμφωνώ μαζί σας πρέπει να καταπολεμήσουμε την καταχρηστική χρήση των αντιβιωτικών. Δηλαδή απλώς ε, το να χορηγούμε ε, αντιβιωτικά στα ζώα ε, για προληπτικούς λόγους είναι κάτι λάθος και νομίζω ότι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στον τομέα αυτή η πρακτική. Σε ό,τι αφορά τώρα το βοηό κρέας και την εισαγωγή από την Βραζιλία. Ξέρετε, εδώ και λίγο καιρό έχω να λάβω τα καθηκοντά μου και το ακούω συνέχεια το ζήτημα αυτό. Οι πληροφορίε που λαμβάνω από τη δική μου υπηρεσία είναι ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τις εισαγωγές, όλες τις εισαγωγές, οποιοδήποτε μου στην Ευρώπη θέλουμε να είναι ασφαλής. Ε, δηλαδή θέλουμε να προέρχεται από από εργοστάσια, σφαγεία που να είναι πιστοποιημένα από το αρμόδιο κτηνοτρικό μας γραφείο. Ξέρετε ότι οι πληροφορίες που είχα σε σχέση με τη Βραζιλία είναι ότι από τα 10.000 ε, μονάδες που ε, εξάγουν στην Ευρώπη σήμερα μόνο 1936 νομίζω τελικά εξάγουν στην Ευρώπη γιατί έχουν το καταλληλοπιστοποιητικό. πιστοποιητικό. Άκουσε τι υπόθηκε εδώ για την Μπερκοσούρ, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και φυσικά θα συζητήσω το θέμα αυτό και φυσικά θα παρουσιάσω και τις ανησυχίες των καταναλωτών και τις ανησυχίες της ασφάλειας των τροφίμων αλλά και των γεωργών. Θα πρέπει να κάνω μια δήλωση ότι η Ευρώπη επιμένει στο ότι θέλουμε να έχουμε τόσα καλά πρότυπα για τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία να συνάδουν με τα ίδια προϊόντα που απαιτούμε τους, με πρότυπα που απαιτούμε από τους δικούς μας παραγωγούς. Δηλαδή δεν προβαίνουμε σε εισαγωγές απλώς για να ικανοποιήσουμε τους εξαγωγείς. Φυσικά, ανάλογα πρότυπα ζητάμε να γίνουν σεβαστά και από τους δικούς μας παραγωγούς ε, για να γίνει σεβαστή και η νομοθεσία αλλά και για να είμαστε και σίγουροι ότι υπάρχει προστασία και στον τομέα της κτηνοτροφίας και όχι ότι απλώς έχουμε ένα τελικό προϊόν το οποίο χαίρει προστασίας και πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο την ποιότητα ε, των τροφίμων που έρχονται στο τραπέζι μας, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε και το μέλλον του όλου τομέα. Τώρα για τη σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια των βοηθών, ε, φυσικά το εξετάζουμε το θέμα αυτό. και μπορώ να σας πω ότι θα υπάρξει κάποια χαλάρωση των ε, σημερινών απαιτήσεων. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δεσμευτώ για το επίπεδο αυτής της ε, χαλάρωσης που θα επέλθει, αλλά καθώς το θέμα της πογκοδούς εγκεφαλοπάθειας ε, των βοηθών έχει τεθεί υπό έλεγχο και αυτό χάρη στη δράση που έχει αναλυθεί στο παρελθόν, πιστεύουμε ότι μπορούμε να μην είμαστε πλέον τόσο αυστηροί, χωρίς φυσικά από την άλλη να θέτουμε σε κίνδυνο την ποιότητα, γιατί δεν θέλαμε να ανακύψει εκ νέου μια τέτοια κρίση όπως αυτή που βιώσαμε στο παρελθόν. Ελπίζω να κάλυψα όλα τα ερωτήματα που ακούστηκαν. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα έχετε και την ευκαιρία να επανέλθετε, αλλά σας ευχαριστώ και για κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, που κάνατε. Δηλαδή το να συνδέετε την ευημερία των ζώων, ε, με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους γαματαφομίκρων. Εδώ υπάρχουν ε, αρκετές ευαισθησίες. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα αυτό και σημαντικό αλλά εγώ πιστεύω ότι το να ακούσουμε περισσότερο την επιστήμη ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κάνουμε σοβαρές επιλογές. Ας ε, ξαναμπούμε τώρα και πάλι στη συζήτηση. Σας ε, παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο, γιατί δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα στη μυρση διάταξη. Αντετές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που εμφανίζεστε τόσο νωρίς στη θητεία σας <clears throat> εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας. Ως εκπρόσωπος των βουλευτών της πολιτικής μου που ασχολούμαστε με τη Γεωργία, θα ήθελα να σας πω ότι χρειάζεται πλήρη συνεργασία με τους αγρότες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, όπου ένας, ε, μάθαμε ότι ένας γεωργός είχε φτιάξει οικειοθελώς ένα φράχτη το από θάμνους ή από δέντρα και εμφανίστηκε μετά ο, Γεωργό, ο, ο Υπουργός από το κόμμα των Πρασίνων και είπε προσοχή 15 μέτρα δικαιούστε μόνον να ε, φυτέψετε μακριά από τέτοιους ε, ε, φράχτες. Αυτό σημαίνει καταδίκη βέβαια της, ε, των ε, φραχτών αυτών. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία. Σήμερα υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν διατηρήσει τα κτήματά τους επί εκατονταετίες ε, μέσα στις οικογένειες αυτές. Και πάμε τώρα να τα προστατεύσουμε εμείς. Ας το σκεφτόμαστε όταν ερχόμαστε να χαρακτηρίζουμε περιοχές ως υποπροστασία. Και σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε σχετικά δηλαδή με τις εισαγωγές τροφίμων ότι αυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις δικές μας προδιαγραφές. Έχω επισκεφθεί πολλές χώρες και πάντοτε αγανακτώ όταν διαπιστώνω ότι επιβάλλουμε στους Ευρωπαίους αγρότες αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες. Και πριν κύριε Επίτροπε τώρα αν αρχίσετε να σκέφτεστε και άλλα μέτρα για την μεταφορά των ζώων, σκεφτείτε λιγάκι ορισμένες χώρες όπως την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ταϊλάνδη και την Αυστραλία και πώς αυτές μεταφέρουν τα ζώα τους. Συλλέξτε εμπειρίες από τις χώρες αυτές και ελάτε να τις συζητήσετε ξανά μαζί μας είναι σημαντικό και οι χώρες αυτές να τηρούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές. Εν τέλει, ένα θέμα το οποίο στη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, τη Βαβαρία, παίζει σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν στη Βαβαρία πολλές μικρές λίμνες όπου υπάρχουν ψάρια. Ε, οι Κυπρίνοι, ψάρια του γλυκού νερού. Έρχονται λοιπόν πουλιά τα οποία ψαρεύουν μέσα στις λίμνες αυτές και τις αδειάζουν. Και τώρα ερχόμαστε εμείς να τα προστατεύσουμε τα πουλιά αυτά. Με, μου τηλεφώνησε σήμερα το πρωί ένας αγρότης ο οποίος προετών είχε βάλει 20.000 ψάρια στη λίμνη του. Του έχουν μείνει 500. Αν δεν βρούμε λύση για το πρόβλημα αυτό δεν θα ξαναβάλει ψάρια στη λίμνη του ο αγρότης αυτός. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα γιατί οι λίμνες αυτές πρέπει να διατηρηθούν, πρέπει να είναι ζωντανέ. Έχουμε στην Ευρώπη τώρα παραπάνω από ένα εκατομμύριο κόρμοράνους, περί αυτών των πουλιών πρόκειται, οι οποίοι έρχονται και αδειάζουν τις λίμνες. Κάποτε επιβάλαμε την προστασία αυτή γιατί είχαμε μοναχά 7.000 ζευγάρια κορμοράνων τα οποία ε, έφτιαχναν φωλιέ και αναπαράγονταν. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, χρειάζεται άλλη ρύθμιση. Μάρτιν Ερώτηση προς τον Επίτροπο Αρμόδιο για την Προστασία του Καταναλωτού. Μέχρι τώρα δεν έχουν ικανοποιήσει οι απαντήσεις σας που λέτε ότι σχετικά με την γενετικά τροποποιημένη πατάτα αμφλόρα δεν υπάρχει θέμα συμβίωσης με άλλα ε, θετικά προϊόντα. Πήγα τώρα και πρόσφατα και ρώτησα και μου είπαν ότι μένουν πολλοί βολβοί μέσα στην ε, γη μετά από την ε, εσοδεία της πατάτας. Και η πατάτα είναι πολύ σημαντική και η διατροφή του ανθρώπου. Ήδη βρίσκεται στην τέταρτη θέση σημασίας. Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχετε σωστά αξιολογήσει τα θέματα και για παράδειγμα αναφέρομαι στα, στην αντοχή στα αντιβιωτικά. ούτε είναι και σαφές για μας γιατί ως αρμόδιο στην προστασία των καταναλωτών δεν βάζεται πιο πολύ στο προσκήνιο της ανάγκης προστασίας του καταναλωτού. Λέτε κάθε φορά ότι πρέπει να ζυγίσει κανείς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της γενετικής τροποποίησης. Μετά όμως μέμφεστε του αντίθετου με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς λέγοντα ότι είναι δήθεν παρασύρονται από το συνέστημα. Δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές και πρέπει να ακούσετε και τα επιχειρήματα αυτών που είναι αντίθετοι. Τώρα έρχομαι σε θέματα σπόρων. Υπάρχει ρύθμιση τώρα μηδενική ανοχής. Όταν λέτε τώρα όμως ότι οι σπόροι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι στο μέλλον από οποιαδήποτε γενετική τροποποίηση, αυτό έχει βέβαια μεγάλη σημασία. Και ένα ερώτημα τώρα σχετικά με την κλωνοποίηση. Σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή αργότερα θα ταχθείτε υπέρ του να ρυθμιστεί η κλωνοποίηση μέσα στον κανονισμό Novel Food. Είπατε ότι θα αναμείνετε πρώτα μια μελέτη και μετά θα μπορέσετε να λάβετε την απόφασή σας. Τώρα, εφόσον πρόκειται για ρύθμιση μέσα στα πλαίσια του Novel Food και αντίθετα με τα όσα ζητεί το Κοινοβούλιο, γιατί το Κοινοβούλιο για το θέμα της κλωνοποίησης είπε καθαρά και εξάστερα οτι ότι πρώτα-πρώτα θέλουμε επιβολή απαγόρευση της εισαγωγής και μετά λήψη απόφασης μέσα στη διαδικασία συναπόφασης. Γιατί δεν περιμένετε λοιπόν πρώτα να γίνει αυτό, γιατί δεν καταθέτεται πρώτα σχέδιο νόμου και να προχωρήσει με τον τρόπο αυτό. Γιατί πάτε τώρα να τα ρυθμίσετε μέσα του κανονισμού Novel Food, δημιουργώντας έτσι τελεσμένα γεγονότα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάρκιν. Η κυρία Χάρκιν. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσία του εδώ. Καταρχήν, να σας ρωτήσω για την χαμηλή παρουσία του G-Mount των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε διάφορα τρόφιμα. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει από πολλές χώρες ε, προϊόντα σόγιας ε, και ε, είναι κυρίως εκεί παρόντες οι γενετικοί τροποποιημένοι οργανισμοί μας είπατε ότι η απαγόρευση δεν θα εξυπηρετούσε κανέναν. Ε, όμως, κοιτάξτε, εδώ ε, βλέπουμε ότι οι ανησυχίες ε, και επισημάνσεις αυξάνονται. Είναι πρακτικό πρόβλημα και αφορά το θέμα του χρόνου και της αποτελεσματικότητας. Τι προτείνετε να γίνει με το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω, το έθεσαν ε, και άλλοι συνάδελφοι, θα είμαι σύντομη, μιλήσατε για την αξιολόγηση για το κόστος τους γιοργούς και θέλετε να έχετε μια ε, ε, συνολική εικόνα για το κόστος της νομοθεσίας. Το απόγευμα θα συζητήσουμε ε, το θέμα του αξιοπρεπού στο δίκαιο εισοδήματο ε, για τους γεωργούς. Η Κομισιόν είπε από το 1995 στο 2005. Αν ε, δούμε την ευρωπαϊκή προστομένη αξία που, προτε... που προστέθηκε στην διατροφική αλυσίδα, η μόνη πραγματικά προστέμενη αξία ήταν στο γεωργικό τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία στενή σχέση μεταξύ των δύο επιτροπών ε, Γεωργίας και Περιβάλλοντος όταν θα εξεταστεί το θέμα αυτό. Δηλαδή πολλές φορές ε, κάθε μία επιτροπή έχει μία μεμονωμένη ε, εικόνα και δεν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος στους αγρότες. Κύριος Γιάλεφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κύριε Επίτροπε. Σημαντικά θέματα τονίσατε και χρειάζεται βέβαια και μια καλύτερη διασύνδεση των διαφόρων πόρων που διαθέτουμε. Τώρα, πρώτα, για τα, για τα αντιβιωτικά. Εάν κατάλαβα καλά, η χρήση αντιβιωτικών για πάχυνση των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται. Αυτό είναι σαφές. Αντιβιωτικά χρησιμοποιούνται πλέον ε, σε μεμονωμένο ζώο και εφόσον αυτό παρουσιάζει κάποια ασθένεια. Άρα εδώ χρειάζεται προσοχή διότι με τέτοια λόγια ε, οδηγούμε σε ασφάλεια τον ε, καταναλωτή. Οι περισσότεροι αγρότε, τουλάχιστον στη δική μου εκλογική περιφέρεια και στη Γερμανία γενικότερα, δεν χρησιμοποιούν αντιβιωτικά ούτε για πάχυνση και εφόσον χρησιμοποιούν αντιβιωτικά, αυτό είναι μονάχα σε μεμονωμένα ζώα και μόνο για του λόγου είπα. Δεύτερο, Χάρηκα που άκουσα να λέτε ότι θέλουμε να παίξουμε και ρόλο πρωτοπόρου για προστασία των ε, φυτών και των ζώων κτλ. Αλλά εάν ήμουν στη θέση σας θα προσπαθούσα να συμβάλλω ώστε και στις εισαγωγές να ισχύσουν οι ίδιες προδιαγραφές. Εσείς θα δείτε πλήρη υποστήριξη από εμά εφόσον αναλάβετε παρόμοιε νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Διότι ο καταναλωτή έχει εν τέλει το δίκαιο όταν αγοράζει το δικαίωμα, δηλαδή όταν έχει αγοράζει, όταν αγοράζει μάλλον εισαγόμενα προϊόντα να γνωρίζει ότι έχουν παραχθεί με τρόπο παρόμοιο όπως με αυτόν που ε, ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ενώ δηλαδή από άποψη ασφάλεια. Ίσως έχουμε λάβει ορισμένε αποφάσει που δεν ήταν απόλυτα σωστέ. Και μιλώ ιδιαίτερα για την υγιεινή και μεταφορά των ζώων. Στη Γερμανία έχουμε πολλά μικρά κρεοπολία τα οποία είχαν το δικαίωμα μέχρι τώρα να προβαίνουν σε σφαγή ε, τα ίδια. Τώρα όμω οι προδιαγραφέ υγιεινής είναι πια τόσο υψηλές που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές μονάχα τα μεγάλα σφαγεία. Άρα τότε τα ζώα πρέπει να μεταφερθούν μέχρι τα σφαγεία αυτά. Λοιπόν, για σκεφτείτε λιγάκι τώρα ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ δύο στόχων. Εμένα με ενοχλεί, γιατί εγώ ασχολούμαι στην πράξη με την γεωργία, διότι δεν μπορώ να σφάξω το ζώο το οποίο το έχω μπροστά μου και χρειάζεται να μεταφέρω το ζώο 50 χιλιόμετρα μέχρι το επόμενο σφαγείο. Ίσως υπάρξει ε, δυνατότητα να τα αποφύγουμε τις αντιφάσει αυτές εφόσον καταλήξουμε σε κάποιες ορθές συμβαστικέ λύσεις. Αυτά, αυτά ήθελα να πω. Μετά θα, από ε, τον τωρινό μιλητή ο κύριος Δανέλη θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. ο, ο κ. Γκλάτφελτερ. Έχω γράψει μια σχετική επιστολή. Παρ' όλα αυτά θα σας μιλήσω τώρα και όλα σας τα πω και προφορικά. Δηλαδή πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή οι Ουγγρικές αρχές τελευταία βρήκαν προϊόντα φυτικά και ζωικά, δηλαδή κτλ. από ε, χώρες της Ασίας που έχουν κατάλοιπα ζυζανιοκτώνων που φτάνουν μέχρι και εντομοκτώνων που φτάνουν μέχρι και 30 φορές περισσότερα από τα επιτρεπόμενα όρια. Έχουν λοιπόν χημικά κατάλοιπα σε οποροκυπευτικά προϊόντα. Βρήκαν λοιπόν ε, κατάλοιπα ε, χημικών τα οποία απαγορεύεται, των οποίων χρήση απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα έχει απαγορευτεί και η χρήση τους και διεθνώς στη βάση της Συμφωνίας της Στοκχόλμης. Και από το Μαρόκο, για παράδειγμα, το οποίο έχει συνυπογράψει τη σχετική συμφωνία. Και αυτές οι χημικές ουσίες, ακόμα και σε μικρότερες ε, ποσότητες, μπορούν να είναι καρκινογόνες οι ουσίες αυτές τέτοιε περιπτώσει γίνονται όλο και συχνότερε. Στου τελευταίου μήνες σημειώθηκαν 12 τέτοιε περιπτώσει μόνο στην Ουγγαρία. Και πρόκειται για οπωροκυβευτικά προϊόντα κυρίω από, νότιο, από βόρειο βόρειο-αφρικανικέ χώρες όπως το Μαρόκο όπω είπα προηγουμένως καθώ και από χώρε τη Ασία. Χρειαζόμαστε λοιπόν νομικά πλαίσια τα οποία θα επιτρέψουν εξασφάλιση εισαγωγών τροφίμων που να είναι απόλυτα καθαρά. θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κανονισμός 178 ε, του 2000. Έχουν υπάρξει και παλαιότερες τέτοιες περιπτώσεις, όπως τότε που απαγορεύτηκε η εισαγωγή μελιού από την Κίνα γιατί δεν υπήρχαν επαρκείς έλεγχοι που να εγγυώνται την ασφάλεια του προϊόντος αυτού. Θα πρέπει τέτοιοι έλεγχοι τώρα να θεσπιστούν και για τα προιοντα εισαγωγής εισαγωγή βορειοαφρικανικών χωρών καθώς και χωρών της Ασίας. Και παρακαλώ να ζητήσετε από τις υπηρεσίες σας να εξασφαλίσουν την διεξαγωγή σε βάθος ελέγχων και επίσης να προβείται και σε συνεργασία και με τις ενδιαφερόμενες χώρες εξαγωγής, ώστε να υπάρξει κοινή βάση προστασίας του Ευρωπαίου καταναλωτού. Ο κύριος Λεφόλ και μετά ο κύριος Δανέλης. Εγώ δύο παρατηρήσεις θα κάνω πολύ σύντομα για, τις, για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, κύριε Επίτροπε. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ που είμαστε. Θα πρέπει να οργανώσουμε μία συζήτηση που θα ξαναθέτει προς σκέψη την ε, μέθοδο και τις απόψεις για την εξέταση αυτού του ζητήματος. Εγώ θα ήθελα να συναντηθείτε και με τους άλλους ε, πρόεδρους ε, επιτροπών που ασχολούνται με το θέμα, να οργανώσουμε δηλαδή μία συζήτηση που θα θέτει τους όρους για το πώς θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και το θέμα των βιοτεχνολογιών. Δεν μπορούμε να στέλνουμε ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον και να παίρνουμε αποφάσεις όπως αυτή της πατάτας όπου κανένας δεν ξέρει τίποτα. Ξέρουμε ότι για αυτά τα ζητήματα η βιομηχανία πιέζει στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Ευρώπη πιο συγκεκριμένα για την πατάτα. Όλοι άσκησαν πιέσεις. Τώρα εμείς δημοκρατικά πρέπει να βρούμε τα μέσα για να ρυθμίσουμε αυτά τα ζητήματα. Προτείνω λοιπόν σε επίπεδο Κοινοβουλίου και κομισιών να οργανώσουμε επιτέλους μία συζήτηση που θα μας επιτρέψει να κάνουμε επιλογές. Να δούμε τι μπορούμε να δεχθούμε για τη γενετική και για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τι θα πρέπει να απορρίψουμε. Να μην πηγαίνουμε μπαλάκι, δηλαδή μια φορά από την πίεση των των βιομηχάνων και ε, την ε, αντίσταση αυτών που πολύ δικαιολογημένα δηλαδή ε, προσπαθούν να μηνθούν. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Πρόεδρε μια, για πάντα να οργανώσουμε μια συζήτηση. Τώρα για το θέμα των διεθνών ζητημάτων εμπορίου δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι θα εφαρμόσουν τους κανόνες οι άλλοι. Το ξέρετε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι διμερείς συμφωνίες που έχουν συναυθεί στην, Ευρώπη και μερικές χώρες των Άνδεων παραμερίζουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ευημερία και με το περιβάλλον. Εγώ θα έλεγα να δείτε το άρθρο 20 των συμφωνιών του Μερακέσου όπου θα γίνει μία αξιολόγηση των μη εμπορικών κανόνων που θα πρέπει να δεσμευτούμε να εφαρμόσουμε όταν διαπραγματευόμαστε στην ΠΟΕ. Να έχουμε δηλαδή μία σαφή κατευθυντήρια γραμμή να εφαρμόζουμε καθαρά αυτούς τους κανόνες για, που, για τους οποίους μιλάμε όλους, αλλά να μην λέμε ναι, ναι, ναι, ναι, θα τους εφαρμόσουμε όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι κανόνες δεν είναι αμοιβαίοι. Σας παρακαλώ λοιπόν, στα πλαίσια ενός άρθρου που υπάρχει στην ε, ΠΟΕ, να βάλουμε έναν σαφή ε, άξονα για τους ε, κανόνες, τους μη εμπορικού κανόνες. Είναι κοινωνικοί κανόνες και περιβαλλοντικοί κανόνες. Ναι, Στεφάν, συμφωνώ, συμφωνώ στο να γίνει μία ανοιχτή κοσμική συζήτηση για τους μη γενετικά Προπομένως οργανισμούς. Δανέλης. Έλθω στην ε, πρόσφατη πολυζητημένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια άλλη όμως οπτική γωνία. Ε, η απόφαση αυτή πέρα από την αδιαφάνεια που τη συνόδευσε νομίζω ότι αναδεικνύει και κάποιες σημαντικές αντιφάσεις. Δεν θα επιχειρηματολογήσω γιατί είμαι κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και της καλλιέργειάς τους. Θα σταθώ όμως σε δύο κοινέ παραδοχές Πρώτο, στι αρνητικέ επιπτώσει που έχουν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στην βιοπικιλότητα και δεύτερο, στην τρέχουσα πολιτική σήμανση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Στην πρώτη περίπτωση, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβεβαιώσει την προτεραιότητα που δίνει στην προστασία της βιοπικιλότητας έναντι της εντατικοποίησης της γεωργικής παραγωγής, με το πρόσχημα βεβαίως της επιστημιστικής ασφάλειας και πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δίνει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα όρια μεταξύ αφενός της επιδίωξης των στόχων της επιστημιστικής ασφάλειας και της μείωσης του κόστους της παραγωγής και αφετέρου της σημαντικής ε, προτεραιότητάς μας, της προστασίας δηλαδή της βιοποικιλότητας. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει η Επιτροπή να ξεκαθαρίσει με ποια κριτήρια διαμορφώνει την πολιτική ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Με βάση την προστασία του καταναλωτή ή την εξυπηρέτηση εμπορικών συμφερόντων. Διότι αν πράγματι δίνει προτεραιότητα στην προστασία του καταναλωτή, ίσως θα έπρεπε να συμπεριλάβει στα κριτήρια για τη διαμόρφωση της πολιτικής ποιότητας και αυτό το κριτήριο, το δικαίωμα δηλαδή του καταναλωτή, να κρίνει ο ίδιος κατά πόσο διασφαλίζεται η υγεία του ή ακόμα και οι ηθικές του αξίες με την κατανάλωση ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Και βέβαια να αλλάξει την πολιτική σήμανση τροφίμων και γεωρικών προϊόντων αναλόγως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Δανέλη. Ο Τζέιμς Νίκολσον. Μετά ο Νικολέστουκου και μετά τελειώσαμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια σχόλια και μια ερώτηση έχω να κάνω. Σωστά μιλήσατε, κύριε Επιτροπή, για την γραφειοκρατία. Δεν θα ήταν καλή ιδέα κάθε φορά που ψηφίζουμε ένα κανονισμό να καταργούμε και ένα κανονισμό ο οποίος είναι πεπερασμένος. Γιατί ε, νομίζω ότι αυτό είναι μία από τις δυσκολίες ε, ε, που προκύπτει, γιατί πολλές φορές ε, δυσκολευόμαστε στην εφαρμογή μιας οδηγίας, ότι τα διάφορα κρατημένη την εφαρμόζουμε διαφορετικό τρόπο και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και παρακολούθηση από τις Βρυξέλλες ότι υπάρχει ορθή εφαρμογή παντού. Άκουσα τα σχολιά σας ε, ότι υπάρχουν τώρα 1936 εκμεταλλεύσει στη Βραζιλία ε, που έχουν άδεια για να εξάγουν βοιοκρέα στην Ευρώπη. Ενδιαφέρον είναι αυτό και μας είπατε για τους αυστηρούς ελέγχους που έχετε, αλλά πριν ε, από σας ε, ε, οι σας μας είπαν ότι 10.000 εκμεταλλεύσεις ήταν διαπιστευμένες. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την ιστορική κατάσταση και μας ανησυχεί κάπως το θέμα αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε με αρκετό ενδιαφέρον. Άκουσα τα σχόλιά σας για τους γαματαφόμικρων. Πρέπει να βασιστούμε στην επιστήμη. Ε, και άκουσα ότι είπατε ότι πρέπει να συζητήσουμε τις ΗΠΑ γιατί πρέπει να έχουμε ε, μια στρατηγική εικόνα για το θέμα αυτό. Και έρχομαι στην ερώτησή μου ε, σε ό,τι αφορά στο τι θα γίνει το 2012. Δεν είναι εδώ συνάδελφος σήμερα. Αλλά εσείς επιβεβαιώσατε πρόσφατα στην Κομισιόν ότι η απαγόρευση του 2012 θα προχωρήσει. Εντάξει, μάλιστα, γιατί η βιομηχανία εκείνη τη στιγμή αναδιαρθρώνεται, αυτή τη στιγμή αναδιαρθρώνεται προς αυτό και πάρα πολλές εκμεταλλεύσεις πουλερικών ε, ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ για να διαρθρώσουν τη βιομηχανία για να είναι έτοιμη για την κατάσταση αυτή. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι νομίζω και εδώ πρέπει να είμαστε σαφές, σαφείς ότι το 2012 δεν θα δώσετε παρέκκληση ότι θα σεβαστείτε τη δέσμευσή σας, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επενδύσεις που γίνονται, ότι δεν θα υπάρχει επέκταση και δεν θα υπάρχει χαλάρωση της κατάστασης. Και επίσης ε, να σας πω και το εξής, νομίζω ότι πρέπει να δούμε και ποιε είναι οι δυνατότητε μας, γιατί μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση, να μην μπορούμε να ε, προμηθεύουμε το 2012 του καταναλωτέ με τον αριθμό των αυγών που θα θέλουν. Έτσι λοιπόν πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό. Και μετά από όλα τα σχολεία μου θα ήθελα να σα ευχηθώ ε, και καλή έκτιση της θητείας σας. Μάλιστα, ο κ. Λουκουλέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλωσορίσατε κύριε Επίτροπε. Σύμφωνο απόλυτα μαζί σας σχετικά με το σημαντικό ρόλο της ε, καινοτομίας και της πρόοδου στον τομέα της γεωργίας. Φυσικά. Θα πρέπει να ανησυχούμε και με όσα απασχολούν τους καταναλωτές για τη χρήση ορισμένων προϊόντων Μιλήσατε για τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και δεν θα σταθώ σε αυτό το θέμα. Αλλά θα σταθώ στο... Η medium είναι ένα παρασυτοκτόνο του οποίου έχει παραταθεί η χρήση στη Ρουμανία για τρία χρόνια. Και αυτό διότι υπάρχει μία συμφωνία σχετική με την Ένωση. Εγώ δεν θα σταθώ στη χρήση αυτής της ουσίας ε, στη Γεωργία, αλλά θα σας πω ότι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διαφωνούν με τη χρήση αυτού του φυτοφαρμάκου. Τι έχετε να πείτε σχετικά εσείς για τη μεταφορά των ζώων. Εσείς επιμείνατε ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον ισχύοντα κανονισμό και μετά να βρούμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά όσον αφορά στην μεταφορά των βοηδών προς τη Ρουσία, δεν γίνονται σεβαστοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Εμείς προσποιούμαστε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και επίσης η Ρωσία προσποιείται ότι σέβεται τους κανονισμούς μας. Τώρα για τις ε, υψηλές προδιαγραφές ε, ε, επισητιστικής ασφάλειας και ασφάλειας των τροφίμων. Να ξέρετε ότι σε αυτόν τον τομέα οι επιδοτήσεις στους αγρότες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης είναι πολύ μικρότερες. Ισονομία δεν σημαίνει ισότητα πολλές φορές. Τι έχετε να πείτε. Και επίσης, στην ε, Μολδαβία, στη δημοκρατία της ε, Μολδόβα, τι ξέρετε για τις εξαγωγές αρνιών στην Ευρώπη. Ο Λιμάνσκι για ένα Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Σημερίζομαι τη δυσαρέσκεια και τον θυμό του προλαλήσαντος Ούγγρου συναδέλφου. Εμείς στην Ουγγαρία εισάγουμε κυπευτικά τα οποία έχουν λεκέδες ζυζανιοκτώνων δεν είναι μόνο από τη Βόρεια Αφρική που έρχονται όλα αυτά αλλά και από άλλες χώρες, άλλες τρίτες χώρες. Εμείς εισάγουμε τοξικά τρόφιμα και αυτό γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι στις τρίτες χώρες. Τα, τα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ λοιπόν εμπορεύονται στην Ουγγαρία αμφίγινα τρόφιμα. Σκάνδαλο αυτό στην Ουγγαρία και θα σας στείλω και όλη τη σχετική τεκμηρίωση για να το διαπιστώσετε. και όλα αυτά δεν περιορίζονται στις εισαγωγές από τις χώρες της Βορείου Αφρική. Όπως είπε και ο κύριος Λότφελντερ. Υπονοήσατε κύριε Επίτροπε ότι μόνο τα κράτη με, ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προστατευθούν από αυτές τις εισαγωγές. Φυσικά, αν υπάρχει πρόβλημα, σίγουρα δεν θα πρέπει αυτά τα τρόφιμα να πάνε στο τραπέζι των καταναλωτών. Και εδώ μιλάω και για την ε, υγεία των καταναλωτών και για τον κτηνιατρικό τομέα, αλλά αυτά πρέπει να τα ελέγχουν, να τα οι εθνικές αρχές των κρατών μελών. Κύριε Επίτροπε, είναι σημαντικό να προειδοποιήσουμε τους συμπολίτε μας για όλα αυτά, για να καταλάβουν πώς διαρθρώνεται όλο το θέμα των κοινοτικών και εθνικών αρμοδιοτήτων. Ισμάνσκι για ένα λεπτό, ο Επίτροπος πρέπει να φύγει, να τον αφήσουμε λοιπόν να απαντήσει μετά. Ισμάνσκι για ένα λεπτό. Moje <clears throat> pytanie zadaję w imieniu grupy posłów e, e Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξή. Πρόκειται για μια ερώτηση στην οποία απάντησε μη ικανοποιητικά η Κομισιόν. Μιλάτε για το μόνο 810. Σε έξι χώρες απαγορεύτηκε η καλλιέργεια αυτού του υβριδικού καλαμποκιού. Μας είπε η Κομισιόν ότι η απαγόρευση στην Αυστρία και στην Ουγγαρία συνδέεται με την ε, βλαπτικότητα για τη δημόσια υγεία αυτού του καλαμποκιού. Αλλά βλάπτει μόνο τους Ούγγρους και τους Αυστριακούς. Θα έπρεπε να βλάπτει όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν μας είπε ότι εξετάζει τη δυνατότητα λήψης απόφασης ε, σχετικά. Πού βρίσκεται όμως αυτή η απόφαση και τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίζουν ανεξάρτητα αν μπορούν να καλλιεργούν ή όχι γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ολοκληρώσαμε. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε για να απαντήσετε και σε αυτό το δεύτερο μπλοκ ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας Ευχαριστώ επίσης που ακούσατε όλα όσα σας είπαμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, γιατί η αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα μας βοηθήσει όλους μας να πράξουμε το πέλτιστο για τους πολίτες. Και πιστεύω πραγματικά ότι τελικά τους πολίτες πρέπει να έχουμε κατά νου. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα να παρευρίσκομαι εδώ και να ακούω τις διάφορες ε, προτάσεις ε, που μου υποβάλλετε, τις οποίες καλωσορίζω. Τώρα, για να ξεκινήσουμε και πάλι με τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τη διαχείρισή τους. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς θέτουμε τα θέματα αυτά. Καλωσορίζω τα σχόλια που ακούστηκαν, ότι θα πρέπει να έχουμε μία συζήτηση που θα επικεντρώνεται στο θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε απλώς συναισθηματικοί. Και φυσικά μην νομίζετε ότι όλα τόσο είπατε τα αντιμετωπίσω ως συναισθηματικές τοποθετήσεις, αλλά άκουσα κάποια επιχειρημάτα που είναι παραπλανητικά, ακριβώς γιατί διέπονται από το συνέστημα. Δηλαδή όταν κάποιος κάνει μια δήλωση ότι η πατάτα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό διατροφικό προϊόν και δεν θα μετατραπεί σε τύψη. Είναι ένα βιομηχανικό προϊόν ε, και θα μετατραπεί σε άμυλο και αυτό ε, θα εμποδίσει την υλοτόμηση πολλών δέντρων για να δημιουργηθεί στη συνέχεια για να κατασκευαστεί καρτί. Ε, έτσι λοιπόν πρέπει εδώ να έχουμε κατά νου όλες τις πληροφορίες και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια αντικειμενικότατη άποψη, μια πολύ αντικειμενική συζήτηση προκειμένου να μπορέσουμε να συζητήσουμε με βάση τη λογική. Εγώ είμαι υπέρ αυτού, θα το συζητήσουμε αυτό στην Επιτροπή και καλωσορίζω μία συζήτηση μεταξύ των Επιτροπών ε, Γεωργίας και Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό. Και φυσικά θέλω να ακούσω ποια είναι η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτού. Στο παρελθόν έχει τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει παρουσιάσει τους κανόνες στην Κομισιόν. Και εμεί βάσει αυτών των κανόνων τώρα ε, αναλαμβάνουμε δράση. Δεν ε, παραβλέπουμε τους κανόνες αυτούς. Δηλαδή, ούτω ή άλλω, κανεί δεν μου δίνει λευκό επιταγή για να αποφασίσω εγώ όπω θέλω. Δεν ε, πρόκειται εδώ για μία υποκειμενική απόφαση που, μπορεί εγώ, που μπορώ εγώ να λάβω. Πρέπει να λάβω μία αντικειμενική απόφαση βάσει των επιστημονικών πορισμάτων και βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών που μα έχει δώσει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να κάνουμε και πρέπει να επικεντρωθούμε επί των τρόπων με τους οποίους θα καταστήσουμε πιο λεπτομερείς αυτούς τους κανόνες έτσι ώστε να διασκεδαστούν και ανησυχίες. Ακούσαμε και τα σχόλια για τη βιοπικιλότητα και τα Δεν θα σχολιάσω επί των θεμάτων αυτών γιατί δεν είμαι επιστήμονας. Εγώ πρέπει να βασιστώ σε αυτά που μου λένε οι επιστήμονες για τα ζητήματα αυτά. Και γι' αυτό νομίζω ότι τα γεγονότα και μάλιστα τα γεγονότα προκύπτουν από την εμπειρία της καλλιέργειας των γαματαφόμικρων είναι αυτά που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σε αυτά πρέπει να βασιζόμαστε προκειμένου να λάβουμε αποφάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, χαμηλή παρουσία, παρουσία χαμηλού επίπεδου, ναι, καταλαβαίνω τις δυσκολίες ε, του τομέα σε ό,τι αφορά την προμήθεια ζωοτροφών. Κυρίως μιλάμε για πρωτεϊνούχες ζωοτροφέ που δεν ε, παράγουμε στην Ευρώπη. Βασιζόμαστε κυρίως στις εισαγωγές για τις ζωοτροφές και αυτή είναι η πραγματικότητα και στη συζήτηση για, τον, για τους γαματαφόμικρων αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και έχει προκύψει αυτό το ζήτημα επειδή εμείς ως Ευρωπαίοι αντιστεκόμαστε σε ό,τι αφορά τη χαμηλή παρουσία Τώρα εκπονούμε μία πρόταση που θέλουμε να τη φέρουμε εδώ στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση. Πρόταση η οποία αφορά ένα νέο τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούμε αυτή την ε, χαμηλή παρουσία. Φυσικά θα απαιτούνται αξιολογήσεις, αλλά νομίζω θα αλλάξουν ορισμένα ποσοστά ανοχής, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν διακόπτουμε τη ροή ζωοτροφών για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους μας, ε, γιατί τελικά αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος παραγωγής για τους γεωργούς μας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενοχή για τους σπόρους, μηδενική ενοχή, ναι, να σας απαντήσω ότι θα διατηρηθεί. Έλεγχο στις εισαγωγές, άλλο ένα θέμα αποτέθηκε. Έντονα μπορώ να πω ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη να ελέγχουν τα σύνορά τους βάσει των προτύπων που έχουν τεθεί στην Ευρώπη ομοιόμορφα και το ότι αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά με υψηλό ποσοστό ε, φυτογενομικών προϊόντων, σε περιεκτικότητα φυτογενομικών προϊόντων ε, τα βρίσκουμε. Αυτό είναι καλό. Έχουμε και το πρόγραμμα δράσης ε, για τα τρόφιμα και όταν εντοπιστούν προβλήματα με προϊόντα και με προμηθευτές ε, που παράγουν και μας στέλνουν αυτά τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν ε, φυτοφάρμακα απαγορευμένα ή υψηλή περιεκτικότητα σε φυτοφάρμακα, δεν θα τα ανεχόμαστε και θα αναλαμβάνουμε δράση. Τώρα, απαγόρευση κλοβών. Έχω απαντήσει με σαφήνεια, δεν θα υπάρχει επέκταση της παρέκκλησης. Αυτή είναι η απόφαση που έχει ληφθεί από την Κομισιόν και θα διατηρηθεί. Καλωσορίζω το σχόλιο για να διερευνήσουμε το θέμα της ε, παροχής των αυγών και νομίζω ότι θα μπορέσω να είμαι σε θέση να αναφέρω τα νέα στοιχεία εν ευθέτω χρόνο στη δική σας επιτροπή. σε ό,τι αφορά το νεματόδες του πεύκου, δεν σας απάντησα την περασμένη μου ε, παρέμβαση. Εμείς έχουμε εξοδέψει αρκετά εκατομμύρια για να εξαλείψουμε αυτόν τον επιβλαβή οργανισμό που συναντάμε κυρίως στην Πορτογαλία. Θα συνεχίσουμε φυσικά να προσφέρουμε στήριξη στο εγχείρημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε εδώ σήμερα μαζί μας. Ξέρουμε ότι έχετε και συνεδρίαση και πρέπει να φύγετε. Ας κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα για να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Επίτροπο και θα ήθελα όλοι να πάρετε την ε, καρτέλα ψηφοφορίας γιατί, την κάρτα ψηφοφορίας γιατί θα ψηφίσουμε στη συνέχεια. Κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα προς το παρόν.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 σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Έλεγχος από τα κράτη-μέλη της Άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Αυτή η πρόταση θέλει να ρυθμίσει το άρθρο 291 της συνθήκης, δηλαδή τη μετάβαση από την παλιά επιτροπολογία στους νέους κανόνες της Λισαβόνας και που αφορούν στις ε, πράξεις, ε, στις συμπληρωματικές πράξεις. Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει την αυτόματη ευθυγράμμιση της επιτροπολογίας στους νέους κανόνες εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 291 που αποκλείουν εντελώς το Κοινοβούλιο από την αποφασιστική διαδικασία. Υποστηρίζω ότι είναι σημαντικό για τα γεωργικά θέματα η ευθυγράμμιση να γίνεται περίπτωση για να αξιολογούμε πότε υπάρχουν οι όροι για βασικές πράξεις και κατά συνέπεια δυνατότητα του Κοινοβουλίου να παρεμβαίνει στην απόφαση. Εμείς συζητήσαμε για το θέμα αυτό στην προηγούμενη συνεδρίαση και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη προς την πρότασή μου. Θα ψηφίσουμε τώρα αμέσω γιατί η συζήτηση έγινε. Υπάρχει η αντίρρηση. Α, έχουμε μερικές τροπολογίες. Siete tutti pronti per il voto? Είστε έτοιμοι όλοι για να ψηφίσουμε. Έχουμε γρήγορες τροπολογίες. Τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Άλμπερ ζήτησε το λόγο. Α, ε, ε, έδειχνε ότι είσαι υπέρ, ωραία. Το ΕΛΚ είναι υπέρ λοιπόν. Σηκώστε τα χέρια. Κατά. Αποχές. Ωραία. Ομόφωνα. Άρθρο 7. Υπέρ. Κατά. Όμορφο. 8. Υπέρ. Κατά. Ομόφωνα. Το 9 διαγράφτηκε. Πού πάμε, πού πάμε, αλήθεια. Μα γράφει deletion. Α, το 9. Ωραία. Υπέρ το 9. Κατά. Άλλος, έγκριτα. Ομόφωνα. 20. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 10. Υπέρ. Ομόφωνα. Είναι κανείς κατά του άρθρου 10. Άρθρο λέει ο πρόεδρος ενώντας τις τροπολογίες. 11. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές 21 υπέρ κατά αποχές μία αποχή 14 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας 2 υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά αποχές Εγκριντ. Έξι. υπέρ κατά αποχές Τώρα τελική ψηφοφορία για την έκθεση υπέρ κατά κανένας κατά θαύμα θαύμα αποχές Ωραία. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Σας ευχαριστώ όλους. Πάμε στο σημείο 7. Εντολή για τον τριμερή διάλογο για το σχέδιο προπολογισμού του 2011. Μαγκίνες, η την προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν δημοσίευσε το προσχέδιο προπολογισμού. Και η κυρία Μαγκίνες, η συγγήτριά μας, έκανε μια τεράστια προσπάθεια για να αναλύσει όλα τα ποσά ε, που χορηγούνται στο κεφάλαιο Γεωργία και θα μας, δώσει την, θα μας κάνει την ανάλυση τη σχετική. Αλλά πριν δώσω το λόγο στην κυρία Μαγκίνες, να σας πω για τα σχετικά του χρονοδιαγράμματος. Προσέξτε με. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 2 Ιουνίου θα εγκρίνει την έκθεσή της. Έτσι εμείς δεν θα έχουμε το χρόνο να εγκρίνουμε τη γνωμοδότησή μας με την πεπατημένη διαδικασία. Η κυρία Μαγκίνεσε θα στείλει το, τη γνωμοδότησή της στα αγγλικά την επόμενη εβδομάδα. Στις 10 Μαΐου λοιπόν και πρέπει να ορίσουμε 18 Μαΐου την ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών, ούτω ώστε να εγκρίνουμε τη γνωμοδότησή μας 1η Ιουνίου. Πολύ πιθανόν λοιπόν η μετάφραση στις άλλες γλώσσες να μην είναι έτοιμη η μετάφραση για τις 18 Μαΐου. Τα ξαναλέω. Μοιράζουμε το προσχέδιο γνωμοδότησης στις 10 Μαΐου, 18 Μαΐου στις 12 λίγη προθεσμία για την κατάδυση τροπολογιών, εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση 1η Ιουνίου, εγκρίνεται 2 Ιουνίου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και 30 Ιουνίου πάει στον Τρίλογο. Η κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο. Thank you, Chair, and thank you for clarifying the very tight time frame. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ο Επίτροπος Προϋπολογισμών το είπε το μέλλον μετά την κρίση και νομίζω ότι από την δική μας τη σκοπιά είναι σωστό γιατί περάσαμε μεγάλη κρίση. Τα ποσά είναι 2,6 δις και 130 δις για τις, ε, υποχρεω... για τις πληρωμές και υποχρεώσεις. και 44,7% παραπάνω και 41,7% για τις ε, ε, πιστώσεις υποχρεωσίες για τη διαχείριση των φυσικών πόρων που μας απασχολούσαν οι ε, πληρωμές είναι 58 δις και 59,5 δις. Και για τις πληρωμές της αγορές 43,7 δις. Τώρα, το περιθώριο για τον τίτλο 2 για το 2011 είναι 852 εκατομμύρια. Πολύ υψηλότερο από ό,τι προβλεπόταν από προηγούμενες εκτιμήσεις. Αν έρχεται λόγω των ε, προσδοκιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι χαμηλότερες οι πληρωμές για τις ε, αγορές μετά από μια απροσδόκητη βελτίωση που σημειώθηκε εκεί. Και ελπίζουμε ότι όντως έτσι θα γίνει και ιδίω στο γαλακτοκομικό τομέα, όπου περάσαμε, όπω είπα, σημαντική κρίση. Βέβαια, δεν είμαστε βέβαιοι πώ θα ε, εξελιχθεί η αγορά. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για την δημοσιονομική πειθαρχία για το 2011. Το θέμα δεν τίθεται ακόμα. Είχαν υπάρξει κάποιε ανησυχίε, αλλά δεν τίθεται το θέμα για το 2011. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν προκύψει τέτοιο θέμα, θα το γνωρίζουμε, διότι μέχρι την 21η Μαρτίου θα μα το είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω θα δείτε ότι το 2011 δεν σημειώνεται τέτοιο πρόβλημα. Νομίζω ότι ε, το ίδιο θα είναι και το σημειώνω ε, για τους ε, συναδέλφους για το 2010, ότι να αποφύγουμε την δημοσιονομική πειθαρχία. Αλλά πάλι αυτό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των αγορών γεωργικών προϊόντων. Όπως είπε ο ίδιος ο Επίτροπος, πάντως πέρασαν, πέρασαν οι άνετες εκείνες οι μέρες όπου είχαμε μεγάλα περιθώρια στην ΚΑΠ για το 2015 θα υπάρξει ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία. Και το, πρόβλημα, το ερώτημα η περισσότερο δεν είναι εάν, αλλά πόσο. Γιατί θα υπάρξουν και νέες πληρωμές προς τις νέες χώρες μέλη, χωρίς όμως να υπάρξει αντίστοιχη αύξηση του προπολογισμού. Άρα θα γίνουν μειώσεις στις άμεσες πληρωμές για ορισμένες από τις παλαιές χώρες μέλη, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το περιθώριό μας για το 2013. Και αυτό όταν θα έχουμε να συζητήσουμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά και ευαίσθητα για το έργο μας εδώ της Επιτροπής Γεωργίας αλλά και για τους αγρότες. Επίσης για την ΚΑΠ από 42% κατεβαίνουμε κάτω από 40% το 2013 για τώρα μέτρα αγοράς. Μείωση κατά 1 δις για το 2013 και αυτό περιλαμβάνει και 300 εκατομμύρια που, έχουν ε, δοθεί, που δόθηκαν μάλλον στον προπολογισμό του 2010, 300 εκατομμύρια όπως είπα υπέρ του γαλακτοκομικού τομέα. Εάν τα δούμε αυτά μέσα στο πλαίσιο αυτό και τα συγκρίνουμε, συγκρίνουμε τον προπολογισμό 2010 με τον προπολογισμό για τον οποίο μιλάμε το 2011 δηλαδή, οι δαπάνες για την αγορά θα μειωθούν σημαντικά από 7,4% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ σε 5,6% για το 2011. Τονίζω και πάλι ότι αυτά βασίζονται στις προσδοκίες μας σχετικά με το πώς θα κινηθούν οι αγορές και ιδίως αυτή του γαλακτοκομικού τομέα για το 2011. Και πάλι τονίζω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να δούμε ποιες είναι οι απόψεις της Κομισιόν γιατί κανένας δεν μπόρεσε να προβλέψει τις αυξήσεις ή και τις καταρρεύσεις τιμών και για να είμαστε έγκαιρα προετοιμασμένοι, αυτές που ζήσαμε δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι έχουμε διαθέσιμο για το 2011 εφόσον σημειωθεί κάποια κρίση. Και δεν νομίζω ότι κανένας μας ή καμία μας θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια πράγματα ε, και εδώ στο Κοινοβούλιο. Και οι τιμέ των αγροτικών προϊόντων εξακολουθούν να πέφτουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα δίχτυ ασφαλεία για να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα. Τώρα, για το Ταμείο Γάλακτο, για να υπάρξει κάποια σαφήνεια εν προκειμένου εμείς κάναμε επιτυχημένη εκστρατεία υπέρ αυτών των 300 ε, εκατομμυρίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι πρόκειται για ένα εφάπαξ μέτρο για να στηρίξει την αγορά του γάλακτος και ενημερώνω τους συναδέλφους ότι όλες οι ε, χώρες μέλη έχουν δηλαδή δηλώσει πώς θα δώσουν, πώς θα πάνε τα χρήματα αυτά. Μέχρι τώρα μόνο 12 εκατομμύρια έχουν δοθεί σε γαλακτοπαραγωγούς από τα 300 και αναμένω τα σχόλιά σας. Χρειάζεται να συζητήσουμε επίσης και μια σταθερή, μια διαρκή γραμμή κονδύλιο δηλαδή του προπολογισμού για το γαλακτοκομικό τομέα. Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή του διαγνωστικού ελέγχου και για τον προπολογισμό του 2011, υπάρχει μια πρόβλεψη να χρησιμοποιηθούν χρήματα για συγκεκριμένα μέτρα στις ε, χώρες μέλη. 486 εκατομμύρια προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Το άρθρο 68 προβλέπεται ε, δαπάνηση χρημάτων πάλι για συγκεκριμένους σκοπούς στις χώρες μέλη και για το προπολογισμό του 2011 υπάρχει ένα ενδιαφέρον ποσό 91% όλων των άμεσων ενισχύσεων των γεωργών θα αποσυνδεθούν από την παραγωγή ενώ ε, για το τρέχοντα προπολογισμό το ποσό αυτό είναι 85%. Άρα προχωρούμε με την αποσύνδεση. Και υπάρχει και μια αύξηση 638 εκατομμύρια για συνδεδεμένα και αποσυνδεδεμένα για τις άμεσες ενισχύσεις και για άμεσες ε, πληρωμές στις νέες χώρες μέλη. Και όπως είπα, αυτές θα, ε, θα προχωρήσουν σταδιακά μέχρι το 2013 όπου θα εφαρμοστούν απολύτως. Υπάρχει τώρα η υποστήριξη στο 2011 ε, υποστήριξη προγραμμάτων για στερημένα πρόσωπα και νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν οι συνάδελφοί μου στην ενθάρρυνση προς όλες τις χώρες μέλη να συμμετάσχουν σε αυτά. Αυξημένη τώρα και δαπάνηση για το, ε, δαπάνηση για το food scheme και ο προπολογισμό που δίνεται στις χώρες αυτές είναι για την συμμετοχή τους για το σχολικό έτος 2011-2012. Ορισμένες χώρες μέλη θα συμμετάσχουν. άλλε χώρες μέλη έχουν ζητήσει μονάχα ένα μέρος της χρηματοδότηση αυτής και πάλι τα διαθέσιμα χρήματα θα δοθούν σε αυτές οι οποίες συμμετέχουν πλήρως. Υπάρχει και μείωση των δαπανών από 374, 374 σε 343 για τα φυτογεωνομικά προϊόντα. Δεν είμαι θα βέβαιη για το τι θα γίνει σχετικά με τις διάφορες ασθένειες φυτών ή ζώων. Εγώ λοιπόν ε, αμφισβητώ αν πρέπει να γίνει μείωση. Έχουμε διανύμει σημείο σημείωμα σε όλους τους συναδέλφους σχετικά με μέτρα στον τομέα της γεωργίας. Έχω λάβει κάποιες ε, απαντήσεις σχετικά με μια μεταρρύθμιση στο γραφειοκομικό τομέα. Ευχαριστώ να ακούσω και σχόλια άλλων συναδέλφων. Ευχαριστώ τους συναδέλφους του Υπολογισμών αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δύσκολη διαδικασία. Είπε ο πρόεδρος και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ήταν σωστή μέχρι τώρα η ανταλλαγή πληροφοριών και δεν μπορώ να τονίσω επαρκώ την σημασία που έχει το θέμα αυτό και να παρακολουθεί η Επιτροπή μα, όχι μόνο τον προπολογισμό του 2011 αλλά και το τι θα γίνει μέχρι το 2013 διότι θα είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη κυρία από την άποψη του προπολογισμού και πρέπει να είμαστε απολύτω σε φάση με το ό,τι συμβαίνει. Θα σταματήσω εδώ και θα ακούσω τα σχόλια του συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες. Συμφωνούμε απόλυτα επί της αμεγκαιότητας συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Στεφαν Λεφόλ. Παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μαγκίνες ε, για την εργασία της και κυρίως για την ε, παρουσίαση που μας έκανε, αλλά θα ήθελα ε, και εγώ να απευθυνθώ στην Κομισιόν και να πω ότι έχουμε κάποια περιθώρια στον προϋπολογισμό του 2011 τα οποία ε, τα συμπεριλαμβάνουμε στα Ταμεία Διαχείρισης ε, των Αγορών. Θέλω να μου πείτε πώς η Κομπισιόν ε, μπορεί να προβλέψει μια τόσο θετική εξέλιξη των ε, γεωργικών αγορών στα μελλοντικά έτη για να αιτιολογήσει τόσο μεγάλη πτώση των πόρων για τη διαχείριση των αγορών κυρία Μαγκίνες ε, μας ε, κάλεσε να σχολιάσουμε ακριβώς το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε αυτό να το αφήσουμε ε, να περάσει έτσι χωρίς να υπάρχει μια πραγματική εξήγηση από την Κομισιόν για να μας πει ε, πού βασίζεται για την λήψη της απόφασης αυτής. Γιατί αν ε, εξακολουθούμε να βλέπουμε η ύφεση σήμερα, οι μηχανισμοί παρέμβασης ε, πού θα βρεθούν. Έτσι λοιπόν ήθελα να το επισημάνω αυτό στην κύριε Μαγκίνε. Στη συζήτηση επίσης που είχαμε στο Στρασβούργο ρώτησα τον Επιτροπό για την χρησιμοποίηση αυτών των εκατομμυρίων για το Ταμείο του Γάλακτος. Μας είπατε ότι χρησιμοποιήθηκαν τα 12 εκατομμύρια. Εγώ νομίζω ότι στο πλαίσιο της Επιτροπής μας θα πρέπει να ζητήσουμε, να ρωτήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει που ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί δεν είναι μικρό το μέγεθος του Ταμείου αυτού. Πρόκειται για ένα τομέα που γνωρίζει δυσκολίες και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς σήμερα χρησιμοποιούνται οι πόροι. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να του τονίσουμε και το θέμα αυτό στη συζήτηση. Όμως πραγματικά εγώ σας επισημαίνω αυτό το θέμα της μείωσης των πόρων που αφορούν τη διαχείριση των αγορών. Ευχαριστώ. Κύριος Γκαρσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μαγκίνες ε, για το έργο της, ε, το οποίο είναι ε, πάρα πολύ σκληρό και μπορώ να πω ότι την πιέζει και ο χρόνος. Είδαμε την κρίση του γεωπιστικού τομέα τα τελευταία χρόνια και ότι οι συνέπειες ε, των ε, διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ ήταν ε, πολύ αρνητικές για τους παραγωγούς και είδαμε πόση δυσκολία έχουμε να ελέγξουν τα κράτη-μέλη, τα κοινοτικά σύνορα. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή εμείς στο Κοινοβουλίο να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος εδώ στην Επιτροπή μας. Γι' αυτό προτείνω το εξή να προετοιμάσουμε τις μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής και όταν πετούμε να προωθηθεί η κοινοτική παραγωγή έναντι τρίτων χωρών με την εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος που θα έχει ως ε, στόχο εκστρατείες ε, ενημέρωσης και κατάρτισης στα σημεία πώλησης και επίσης ε, να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή με ενώσει παραγωγών καταναλωτών, με νοικοκυρές έτσι ώστε μέσα από αυτό το πιλωτικό σχέδιο να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και να καταρτήσουμε τους πολίτες για αυτό που θεωρούμε εμείς σημαντικά για να ξέρουν οι τελικοί καταναλωτές τι διαλέγουν στο σούπερ μάρκετ γιατί ένα προϊόν έχει την τάδε τιμή και ένα προϊόν μια άλλη τιμή. Αν συμφωνείτε, μέσω από αυτού του πιλωτικού σχεδίου θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε μελλοντικέ εργασίε έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει τελικά να θέσει εφαρμογή μια εκστρατεία σε κοινοτικό επίπεδο. Να εξηγούμε τις, ε, τα πρότυπα ποιότητα διατροφική ασφάλεια, να εξηγούμε σε τη συνιστατή ευημερία των ζώων, ε, τα περιβαλλοντικά μέτρα προστασία του περιβάλλοντο Επίση, να εξηγούμε πώ μπορούμε να προστατεύσουμε ε, τον παραγωγό αλλά και τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε περισσότερε πληροφορίε έτσι. Θα αυξήσουμε την ελευθερία ε, του καταναλωτή και το σύστημά μα θα είναι πολύ πιο διαφανέ και δημοκρατικό. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτό το προτείνω εδώ. Ελπίζω να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε και να κατορθώσουμε επίσης ε, να αναδείξουμε τις ε, προσπάθειες που καταβάλει η Επιτροπή με το λογότυπο λόγου χάρη που έχουμε θετήσει και που θα θέσουμε σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Ευχαριστώ την κυρία Γαρσία Νικουλέσκου και μετά Κάπουλο Σάντος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την κυρία Μαγκίνες για την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ που ζητήσατε συγκεκριμένα σχόλια από εμά σε ό,τι αφορά αυτό το πιλωτικό σχέδιο. Θα ήθελα και εγώ να προτείνω ένα πιλωτικό σχέδιο με τη σειρά μου. Ε, να έχουμε ένα πρόγραμμα είδους εράσμους για τους νέους ε, παραγωγούς. Θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε από το πρόγραμμα Εράσμους για τους νέους επιχειρηματίες, όπως και οι νέοι επιχειρηματίες και οι νέοι γεωργοί θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα ε, και θα μπορούσαν ε, να ε, γνωρίζουν μέσω αυτών των ανταλλαγών ποιες είναι οι βαλιστικές πρακτικές. Το έχω συζητήσει αυτό με την κυρία Γκαρτσία, με τον κύριο Τζόμπαρτη. Θέλουμε μία γραπτή δήλωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα και θα ήταν καλό αν μπορούσατε να υπογράψετε τη δήλωση αυτή. Ευχαριστώ. Λουίς, έχεις το λόγο. Πρόεδρε, η δική μου παρέμβαση ακριβώς ήθελα να φερθεί στα ίδια στοιχεία που ακούστηκαν από το συνάδελφο. Έτσι λοιπόν και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την ιδιαίτερα αισιόδοξη πρόβλεψη της εξέλιξης των αγορών. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να μας δώσει μια εξήγηση προς αυτή την κατεύθυνση. Σικυρίσκη και κατόπιν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριο Σιλό. Σχετικά με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Τι θα γίνει, θα δοθεί η σχετική επιταγή. Εγώ θα έλεγα να δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Κριστίν Πόρτμαν, την εκπρόσωπο της Κομισιόν, και μετά να ξανακούσουμε την κυρία Μαγκίνες, η εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την κυρία Μαγκίνες. Νομίζω μάλιστα και η ακρόαση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα ε, ήταν χρήσιμη. Πρώτα ήθελα να πω ότι σήμερα που διεξάγεται η συνεδρία αυτή, στείλαμε και στην Επιτροπή Γεωργίας και στην Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών το έγγραφο για τον προϋπολογισμό 2011 που συνήθως στέλνουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Επομένως έχουμε τώρα και ε, φέτος επειδή είναι οι νέες ε, αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό στέλνουμε αυτά τα στοιχεία που έχουν και ε, όλα τα δεδομένα, τα ποσά και τα ποσοστά, τα οποία μας οδηγούν στα συμπεράσματα που έχουμε καταλήξει. Το πιο σημαντικό για σας είναι οι προσδοκίες σχετικά με την εξέλιξη των αγορών και γιατί η Κομισιόν ε, καταλήγει σε ένα προπολογισμό που, όπω τονίσατε ορισμένοι εξημών, είναι σημαντικά χαμηλότερος από το περσινό. Είναι σωστό αυτό. Και ο λόγος είναι ότι ο προϋπολογισμός είναι όντως 840 εκατομμύρια λιγότερο, 804 λιγότερο και από αυτά 80 για το γαλακτοκομικό τομέα και 80 εκατομμύρια είναι για το σχολικό γάλα. Διότι όταν συνέτασε ε, ε το σχέδιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπήρχαν επιστροφές εξαγωγών, επιδοτήσει εξαγωγών δηλαδή για το γαλακτοκομικό τομέα, ούτε και άλλα μέτρα τα οποία ε, παρέτειναν την ε, περίοδο παρεμβάσεως πέρσι. Αυτές είναι οι προσδοκίες της Κομισιόν και είμαι βέβαια ότι θα έχετε προσέξει κι εσείς ότι οι γαλακτοκομικές αγορές είναι πολύ διαφορετικές φέτος από όταν πέρσι. Τώρα, σχετικά με το τι θα γίνει. Υπάρχει ακόμα η τροποποιητική επιστολή ε, τη Γεωργίας και έχει την πρόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια τροποποιητική επιστολή για την Γεωργία που θα γίνει φέτος τον Οκτώβριο και θα εξετάσουμε εάν υπήρξε κάποια εξέλιξη σε κάποια αγορά μεταξύ αυτών και των Δημητριακών στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος ε, ε, Λεφόλ αυτό είναι το ένα. Τώρα, δεύτερο, υπάρχει ένα περιθώριο στην, στον υπότιτλο 790 εκατομμυρίων για τα δημητριακά δηλαδή. Μπορεί να έρθει μετά βέβαια από την τροποποιητική επιστολή. Υπάρχει πάντως το περιθώριο αυτό και είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τροποποιητικό προϋπολογισμό εφόσον αυτό ε, ε χρειαστεί ε, για οποιοδήποτε περιθώριο θα παραμείνει μετά από τις αποφάσεις της αρχής του προϋπολογισμού. Τώρα, για το Ταμείο Γάλακτος. Όντως, από 31 Μαρτίου μόνο δύο χώρες έχουν καταβάλει πληρωμές και αυτέ δηλώθηκαν στι 30 Απριλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά η 31 Μαρτίου ήταν και η ημερομηνία μέχρι την οποία έπρεπε οι χώρε μέλη να ειδοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι προτίθεται να κάνουν. Η προθεσμία καταβολή όμω είναι μέχρι 30 Ιουνίου και αναμένουμε βέβαια τα νούμερα που θα μας δοθούν για Απρίλιο, ε, Μάιο και Ιούνιο όπου θα είναι για ε, τα, ποσά αυτά των 20 εκατομμυρίων που υποτίθεται ότι θα καταβληθούν. θα περιμένουμε να ε, ειδοποιήσουν, να ανακοινώσουν οι χώρες μέλη ε, τι θα κάνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους επόμενους μήνες θα δούμε τι θα κάνουν. Εκεί βρισκόμαστε για το Ταμείο Γάλακτος και για τις προσδοκίες σχετικά με την αγορά. Σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, νομίζω θα τα αφήσω να τα συζητήσετε εσείς. Ευχαριστώ. Μαγκίνης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη κατόπιν των εξηγήσεων της Κομισιόν. Αλλά θα ήθελα η Κομισιόν να καταγράψει τις ανησυχίες αυτής της Επιτροπής σε σχέση με την ουσιοδοξία για τις εξέλιξεις στην αγορά. Και εμείς θέλουμε να είμαστε αισιοδοξοί, αλλά θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστές. Και από ό,τι καταλαβαίνω, το πραγματικό περιθώριο είναι μόνο 400 εκατομμύρια σε περίπτωση κρίσης. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να επικεντρωθούμε σε μικρό ποσό ε, που θα είναι διαθέσιμο αν προκύψει κρίση και πάλι θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κομισιόν για τις εξηγήσεις, ε, όμως ε, μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα πρέπει να καταβληθούν τα ποσά για το Ταμείο Γάλακτος. Τώρα αν μπει σε κρίση αγορά τότε θα χρειαστούν αμέσως πόρους Γεωργία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα των ενισχύσεων. Τώρα για τα πιλωτικά προγράμματα θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους που παρουσίασαν προτάσεις. Αν μπορείτε στείλετε ένα email κατευθείαν. Σας ευχαριστώ για τις ιδέες σας ε, για το πρόγραμμα είδους Εράσμους ε, φαίνεται ότι είναι καλή ιδέα και θα να προσπαθήσουμε να δώσουμε καλύτερες ε, πληροφορίες στους καταναλωτές για τα προϊόντα και τα πρότυπα φαίνεται κάτι λογικό και πάλι ευχαριστώ τους συναδέλφους που συμμετείχαν. Είμαστε ανοιχτοί στο να ακούσουμε καλές ιδέες για πιλωτικά προγράμματα και πάλι να τονίσω στην Κομισιόν την ανησυχία που έχει η δική μας Επιτροπή για τις εξελίξεις των γεωργικών αγορών, για το πώς θα αναπτυχθούν και θα δούμε αν φέτος τον Οκτώβριο θα υπάρξει τροποποιητιστική επιστολή και ευχαριστώ και για την βοήθεια. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ κύριε Μακκίνες. Αν δεν ζητά άλλο το λόγο, μπορείτε να προχωρήσετε έτσι με τον έλεγχο της κατάστασης. Και θα περάσω τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερικής διάταξης που αφορά την ενημέρωση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιτροπολογία για το βιολογικό ίνο. Εδώ να διευκρινίσω ότι σε σχέση με την Επιτροπολογία η Επιτροπή έχει προτείνει τροποποίηση του κανονισμού C889 του 2008 προκειμένου να καθορίσει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού του Συμβουλίου 834-2007 που αφαιρούν συγκεκριμένους κανόνες για το βιολογικό ίνο. Αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Επιτροπή θα ενημερώσει τη δική μας Επιτροπή Γεωργίας για την απόφαση που θα διαθετούταν από τη Διαχειριστική Επιτροπή Ινου 26 ε, Απριλίου για την τροποποίηση του κανονισμού για το βιολογικό ίνο, αλλά η Διαχειριστική Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση. Παρ' όλα αυτά, ε, χαιρόμαστε που βρίσκεται εδώ ο πρόσωπος Κομισιόν που θα μας παρουσιάσει και τη σχετική πρόταση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα γιατί διαφαίνεται πόσο σημαντική είναι η επιτροπολογία στις αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Εμεί ε, ξέρουμε στις περιπτώσεις αυτές και ευχαριστούμε την Κομισιόν για την ενημέρωση που μας έχει δώσει. Ε, θέλουμε να επισημάνουμε ότι μας ενδιαφέρουν αυτές οι πληροφορίες για όλα αυτά τα λεπτά ζητήματα τα οποία συζητούνται σε συνεδριά της επιτροπολογίας. Έτσι λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Ιλό της ΔΕΛΤΑ ΑΓΡΙ για να μας παρουσιάσει την απόφαση. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να σας πληροφορήσω για το προχώρημα των εργασιών σχετικά με την εινοποίηση του βιολογικού σταφυλιού. Ένας ευρωπαϊκός κανόνας ε, συμβατός με τις προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας επιτρέψτε μου να τοποθετήσω στο πλαίσιο της ε, γεωργικής νομοθεσίας αυτό το θέμα. Έχουμε τον κανονισμό 839 του 2007 του Συμβουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές του βιολογικού έχουν ένα κενό. Δηλαδή, η καλλιέργεια του αμπελιού ορίζεται από αυτόν τον κανονισμό, αλλά η εινοποίηση αποκλείεται μέχρι του παρόντος. Εμείς μπορούμε λοιπόν να πιστοποιήσουμε βιολογικά στα φύλλα, αλλά δεν μπορούμε να πιστοποιήσουμε το βιολογικό κρασί. Η μόνη αναφορά που μπορούμε να έχουμε είναι κρασί από βιολογικά στα φύλλα. Αυτό το διαβάζουμε και στις ετικέτες του κρασιού που αγοράζουμε στο εμπόριο. Ο στόχος λοιπόν ορίστηκε από το σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία, το 2004 συμφωνήθηκε αυτό, και ορίστηκε ο στόχος ε, να βρούμε μία προδιαγραφή για την ε, παρασκευή βιολογικού ίνου. Αυτόν τον ε, στόχο τον ε, πετύχαμε κατά τη συζήτηση το 2007 για τον κανονισμό του Συμβουλίου. Ξεκίνησε λοιπόν η Κομισιόν ε, ε, τις εργασίες της, χρηματοδοτώντας καταρχήν ένα σχέδιο έρευνας, το Orwine, τρία χρόνια κράτησε, σε πολλά κράτη-μέλη. Και με πειραματισμούς ε, πάνω από χίλια αγροκτήματα που παράγουν βιολογικό κρασί Αυτές οι έρευνες δώσανε και την επιστημονική βάση και μετά προχωρήσαμε σε ένα σχέδιο κανονισμού το 2009, πέντε φορές το συζητήσαμε αυτό το κείμενο, στην ε, Ρυθμιστική Επιτροπή για τη Βιολογική Γεωργία, που είναι και η αρμόδια επιτροπή για την ε, επεξεργασία αυτού του κανονισμού. Το 2010 η Κομισιόν στις αρχές Απριλίου ενέκρινε μία πρόταση για τους ε, κανόνες βιολογικής συνοποίησης. Η πρόταση βασίστηκε στις ε, συζητήσεις που έγιναν μέχρι τώρα και στα αποτελέσματα του σχεδίου έρευνας. Με, με, λίγα λόγια θα έλεγα ότι βασιζόμαστε στους γενικούς υπάρχοντες κανόνες στην ΚΟΑ κρασιού. Πρόκειται λοιπόν για κρασί, δεν έχουμε καμία παρέκκληση. Κανόνες οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις συνολογικές πρακτικές, ο κανονισμός 666 κάθετος 09 παραμένει στην ισχύ αλλά Ορισμένες ινολογικές πρακτικές δεν επιτρέπονται για τη βιολογική εινοποίηση, διότι θεωρούμε ότι στρεβλώνουν το φυσικό χαρακτήρα του προϊόντος προέλευσης και υπάρχει και μία λίστα ε, ουσιών που επιτρέπονται για την εινοποίηση. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, αυτό το σχέδιο κανονισμού το έχουμε στην ημερήσια διάταξη της Αρμόδιας Επιτροπής. Τον είχαμε καταρχήν στις 26 Απριλίου σε μια πρώτη συνεδρίαση και 18 Μαΐου έχουμε μια δεύτερη συνεδρίαση. Και θα ζητηθεί η γνώμη της Επιτροπής. Υπάρχει στην αναζήτηση πλειοψηφία στα κράτη-μέλη ένα ρίσκο να μην την πετύχουμε αυτή την πλειοψηφία. Διότι ορισμένα θέματα τεχνητού τύπου ε, δεν βρίσκουν σύμφωνα ε, τα κράτη. Το ένα είναι η ανώτατη περιεκτικότητα σουλφίτ θειοδών στο κρασί ορίστηκε μία ανώτατη οροφή που είναι διαφορετική όπως και στην ΚΟΑ δηλαδή από τον ένα τύπο κρασιού στον άλλον, αλλά θα ήταν πολύ χαμηλότερο αυτό το πλαφόν, αυτή η οροφή για τα βιολογικά κρασιά. Από ότι δηλαδή στα συμβατικά κρασιά. Και γύρω σε αυτό το, από αυτό το θέμα υπάρχει διαφωνία. Τώρα, αν δεν πετύχουμε πλειοψηφία στις 18 Μαΐου, η Επιτροπή θα εφαρμόσει την επιτροπολογία έτσι όπως υπάρχει, ισχύει σήμερα και έτσι όπως ορίστηκε στην ε, απόφαση του Συμβουλίου του 1999. Μετά τις 18 Μαΐου λοιπόν και μετά από αρνητική ψηφο η Επιτροπή ε, είναι υποχρεωμένη να υποβάλει την πρότασή της στο Συμβούλιο το Συμβούλιο έχει στη διάθεσή του τρεις μήνες για να αποφασίσει και θα διαβιβάσει φυσικά την πρόταση και ε, προς πληροφόρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλαμε λοιπόν με την παρουσία μας σήμερα να σας πληροφορήσουμε προκαταβολικά για τη διαδικασία στην περίπτωση που έχουμε αρνητική ψήφο. Βέβαια έχει χρόνο, επαρκή χρόνο η Κομισιόν να εγκρίνει μια πρόταση για το βιολογικό κρέσι πριν από, την, ε, από τον τρίγο του 2010 για να μπορέσουν δηλαδή οι βιολογικοί να πιστοποιήσουν έγκαιρα τα κρασιά τους. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Ιλό και την ε, Εκτελεστική Επιτροπή. Ο Χέρμπερτ Ντόρφμαν ζήτησε το λόγο και μετά η κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το βιολογικό κρασί θα ρυθμιστεί. Τέλεια. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν το είπε. Το πρόβλημα είναι τα θεώδη. Και άμα κολλήσουμε εκεί, η πρόταση της Κομισιόν δεν έχει υπόσταση. μιλάει για τα θειώδη επιτροπή, αλλά τα θειώδη δεν έχουν καμία σχέση με το βιολογικό κρασί. πολύ καλά που χρησιμοποιούμε και τα θειώδη και στα βιολογικά κρασιά. Για τη βιολογική καλλιέργεια μπορεί να υπάρξουν προβλήματα το φθινόπωρο που δεν μπορούμε να παρέμβουμε με εντομοκτώνα, οπότε εκεί παρεμβαίνουμε αυξάνοντας την περιεκτικότητα σε θειώδη. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε στην Κομισιόν, δηλαδή τι γίνεται, μειώνουμε ε, τα θειώδη αλλά μπλοκάρουμε και την κατάσταση. Για μένα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την ε, οποία των κρατών μελών. Τώρα για τις ε, θερμοκρασίες προβλέπεται μια σταθεροποίηση των θερμοκρασιών, θερμική δηλαδή σταθεροποίηση χρειάζεται μία θερμοκρασία όπου θα σταματάει η ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Από τεχνικής πλευράς ε, μου φαίνεται παράλογο αυτό. Πρέπει να καταλήξουμε γρήγορα σε μία απόφαση. Ευχαριστώ Χέρμπερτ, η κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην, ε, στο Intergroup για τα κρασιά το συζητήσαμε και με τους επαγγελματίε ε, το θέμα και έστειλα και μια γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν που δεν μου απάντησε ικανοποιητικά. Πρέπει να γίνει σαφές ότι θα πρέπει να μπορούμε να παράγουμε βιολογικό κρασί σε όλες τις συνοπαραγωγικές περιοχές της Ευρώπης και κάθε χρόνο ακόμα και με άσχημα μετεωρολογικά φαινόμενα. Σε όλα τα επίπεδα λοιπόν παραγωγής και το θέμα των θειοδών, αν τα περιορίσουμε, Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτός ο περιορισμός θα οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Διότι αν θέλουμε λιγότερο υψηλές οριακές τιμές, αυτό δεν, εξάλλου δεν ε, προστατεύει τη δημόσια υγεία, η ίσα δηλαδή η ανεπαρκής θείωση του κρασιού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε υγειονομικό επίπεδο. Για να έχουμε λοιπόν την ίδια ποιότητα και την ίδια δυνατότητα αποθήκευσης, τα συμβατικά και τα βιολογικά κρασιά φιώνονται κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν χρειάζεται εναλλακτική, δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα στην ε, θείωση. Και αν η Κομισιόν θελήσει να κάνει αυτό, περάσει αυτό που θέλει να κάνει δηλαδή, θα δημιουργήσει στρέβλωση στον ανταγωνισμό και δεν θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών. Εγώ έχω και τη θέση των επαγγελματιών ε, στα γερμανικά που λένε τα εξής. Ότι τα κρασιά εφόσον δεν θυώνονται θεωρούν ότι αυτό δεν είναι σωστό βήμα. Και ιδίως στο κλίμα της κεντρικής Ευρώπης, το οποίο αλλάζει συχνά και πυκνά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Και μετά, όπως είπε και ο κ. Στόρφμαν προηγουμένως, λέει και ένα δεύτερο πράγμα που τους φαίνεται ακατανόητο, είναι η νέα ρύθμιση που προβλέπει μείωση της χρήσεως θερμότητας στο πολύ 65 βαθμών ενώ η πρακτική είναι σύντομη έκθεση σε θερμοκρασία 87 βαθμών. Υπάρχουν λοιπόν δύο λόγοι για να μην προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση που βαδίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω μάλιστα ότι πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην δημιουργήσουμε νέες ε, στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων ε, περιοχών ε, και μεταξύ των διαφόρων ποικιλιών. όπου υπάρχει, θα δημιουργηθεί πρόβλημα και στην αποθήκευση και θα δημιουργηθεί και πρόβλημα και με τα κρασιά τρίτων χωρών. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα το καταλάβει η Κομισιόν ότι κάνει λάθος. Αν δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις, Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ιλό για να απαντήσει, να πω μερικά πράγματα για τη μέθοδο. Είναι θεμελιώδες ότι αν η Κομισιόν είναι διαθέσιμη με τους τωρινούς κανόνες να έρθει εδώ και να ξαναπαρουσιάσει την πρόταση, να έρθει πριν ληφθεί η απόφαση, γιατί να έρθει εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας να μας παρουσιάσει μία απόφαση που ήδη έχει γίνει δεκτή, δεν αξίζει τον κόπο για τη συνεισφορά δηλαδή που μπορεί να δώσει και το κοινοβούλιο. Σήμερα ήταν καθαρά ευκαιριακό διότι η Διαχειριστική Επιτροπή του Κρασιού δεν αποφάσισε. Οπότε και εμείς συνεισφέραμε με τις ε, τοποθετήσεις των κυρίων Ντόρφμαν και Λούλινγκ. Θα είμαστε λοιπόν με τους τωρινούς κανόνες να υπάρχει μια τέτοια διάθεση για τα πιο σημαντικά τουλάχιστον θέματα αυτής της Επιτροπής. Εμείς ξέρουμε ότι έχουν προβλεφθεί διαχειριστικές επιτροπές ε, για αυτόν τον μήνα που θα αλλάξουν σημαντικά τους κανόνες του Συμβουλίου για τα οπορικηπευτικά. Και θα θέλαμε να ξέρουμε μερικά παραπάνω από αυτά τα οποία έχει κατά νου η Κομισιόν να αποφασίσει, χωρίς βέβαια να έχουμε και κανένα ρόλο επί της ουσίας. Κύριε Υλό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να απαντήσω στις δύο παρεμβάσεις που ακούστηκαν. Να απαντήσω και στα τεχνικά ζητήματα. Σε ό,τι φορά καταρχήν τη θερμοκρασία σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία ή επεξεργασία με θερμότητα γενικά επιτρέπεται για τους συμπατικούς ίνους, χωρίς δηλαδή περιορισμό στη θερμοκρασία, χωρίς όριο. Όμως για το βιολογικό ίνο θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να ορίσουμε ένα όριο για να μην υπάρχει πλήρης ε, στήρωση του προϊόντος ε, έτσι ώστε ο ε, ιδιαίτερος χαρακτήρας ε, του σταφυλιού να μπορεί να λάβει ιδιαίτερη αξία. Η θερμοκρασία προτείνει η Κομισιόν είναι το μέγιστο 65 βαθμών είναι αρκετά υψηλή η θερμοκρασία. Σήμερα την ε, εφαρμόζουν οι περισσότεροι ίνο παραγωγοί και δεν φαίνεται ότι θα θέτει ιδιαίτερο πρόβλημα για την παραγωγή βιολογικού ίνου. Σε ό,τι αφορά τα θειώδη, αυτό το θέμα έχει συζητηθεί ευρέως. Είναι αλήθεια ότι για τους συμβατικούς ίνους εφαρμόζουμε ένα ανώτατο όριο 200 μιλιγκράμμα ανά λίτρο για τον ερυθρό ίνο, τον ξηρό. 200 μιλιγκράμμα ανά λίτρο για το λευκό και το ροζέ ίνο. Για, μπορεί να φτάσει όμως για άλλους μέχρι και τα 400 mg αναλύτρο. Αυτό για τους ε, συμβατικούς ίνους. Όμως ε, η έρευνα έδειξε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ε, η παραγωγή βιολογικού ίνου μπορούσαν να παράξουν κρασί χωρίς να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέγιστα όρια. Αυτό διαπιστώθηκε όχι βάση μικρού δείγματος, αλλά έλαβε χώρα, υλοποιήθηκε μια ευρεία μελέτη σε χίλιε εκμεταλλεύσει. Έτσι λοιπόν, ε, μειώσεις 50-60% ε, είναι δυνατόν ε, να υπάρξουν για αυτούς τους παραγωγού, ακόμη και για όσους βρίσκονται σε μειονεκτούσες περιοχές, δηλαδή προς τη Βόρεια Ευρώπη. Η συζήτηση έδειξε όμως ότι το οριστεί ένα αυστηρό ανώτατο όριο, δηλαδή δραστική μείωση 50%, λόγου χάρη θα μπορούσε να παρουσιάσει πρόβλημα για ορισμένους παραγωγούς που έχουν συνηθίσει λιγότερο στο να χρησιμοποιούν ε, κάποιες τεχνικές ε, ή αν έχουν μια πιο δύσκολη χρονιά. Έτσι λοιπόν, ε, αυτή η μείωση που προτείνεται είναι 33% για το ξηρό ερυθρό ίνο, δηλαδή από τη 250 στα 200 ε, ε, ε, και για το γλυκό ίνο που ξέρετε χρειάζεται μεγαλύτερη σταθεροποίηση, δηλαδή πιο πολλά Η μείωση είναι 30 mg μόλις, δηλαδή έχουμε ίνους όπως το ice wine και θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο ανώριο του 370 mg ένα λίτρο. Αυτό είναι ανώτερο από ό,τι χρειάζεται. Τώρα είναι ρεαλιστικά τα νούμερα αυτά, γιατί άκουσα ότι μπορεί να ακουστούν και κάποιες κριτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φοβόμαστε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Νομίζω ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί δεν πρέπει να φοβούνται αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Είναι εφικτό να παράξει κανείς κάποιο καλό βιολογικό κρασί πιστοποιημένο σεβόμενο σε αυτά τα νότατα όρια. Το δύσκολο θέμα είναι το θέμα του κλίματος. Ο τρισμένες χρονιές ε, υπάρχει ε, πρόβλημα με το κλίμα, είναι κακός ο καιρός ε, και έτσι λοιπόν η Κομισιόν έχει ένα κανόνα ευελιξίας, δηλαδή εκεί όπου έχουμε εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες θα επιτρέπεται ο παραγωγός που βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση σε μια συγκεκριμένη χρονιά να μπορεί να αυξήσει την περιεκτικότητα σε θειώδη μέχρι το ανώτατο όριο που επιτρέπεται για τα συμβατικά κρασιά. Έτσι λοιπόν ε, με την διάταξη αυτή ε, συμπεριμένουμε ότι το σύνολο των Ευρωπαίων παραγωγών που μπορούν να παράξουν ε, ίνο από βιολογικό σταφύλι σήμερα δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερε δυσκολίε με τον κανόνα που προτείνεται από την Κομισιόν. Με αυτό τον κανόνα, μάλιστα, αυτό ο κανόνα όχι απλώ βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία, αλλά έχει υλοποιηθεί και επί τόπου και μπορεί να συγκριθεί και με ιδιωτικά πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες. Αυτά τα ιδιωτικά πρότυπα εφαρμόζονται και στο Νότο αλλά και σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, δηλαδή στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτά τα ιδιωτικά πρότυπα δεν προβλέπουν ανώτερη περιεκτικότητα σε θειώδη από αυτό που προτείνεται από την Κομισιόν. Θα έλεγα μάλιστα ότι απαιτούν πιο αυστηρά πρότυπα από την πρόταση της Κομισιόν. Είναι ρεαλιστική λοιπόν η πρόταση αυτή και θα μας επιτρέψει να ορίσουμε το βιολογικό ίνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο σημείο αυτό θα έλεγα ότι αν δεν ε, θέλει κάποιος άλλος το λόγο μπορούμε να διακόψουμε τις εργασίες μας. Έχουμε σεβαστεί και το χρόνο. Όχι. Κυρία Λούλινγκ ε, θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Μία φράση μόνο με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες συνοποιούς που λένε ότι δεν είναι σωστό αυτό και ότι θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις ανταγωνισμού. τους έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από αυτούς τους ε, γραφειοκράτες της Κομισιόν. Διερωτώ με, εάν, γνωσ... εάν έχουν τη γνώση οι ε, γραφειοκράτες της Κομισιόν, αν έχουν τη γνώση, τη γνώση την οποία έχουν οι νοποιοί και χρειάζεται λοιπόν να προσέξει ιδιαίτερα η Κομισιόν τι πάει να κάνει. Μάλιστα, ευχαριστώ και πάλι κύριε Λούλινγκ. Θα τα ξαναπούμε στις 3 ε, για να συζητήσουμε το, τον επιστηστικό τομέα.